Mes chers Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σας κύριε Βαντενκάπ και τους Διερμηνείς. Χαιρετώ. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα. Τι να κάνουμε έτσι είναι η ζωή. Σχέδιο μερίσια διάταξης μπορεί να εγκριθεί αν δεν έχετε καμία αντίρρηση τα συνοπτικά, ε, τα πρακτικά μάλλον της 19ης και 20 η Ιουνίου θα θεωρηθούν εγκεκριμένα αν δεν διαφωνεί κανείς. Δεν βλέπω να διαφωνεί. Και αρχίζουμε με το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Γενικός Προϋπολογισμός 2018, όλα τα τμήματα. Και θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον εισηγητή μας που δεν ξέρω είναι και παρόν κατά τα άλλα. Μάλιστα. Α, δεν σας έβλεπα, κύριε Τοσενόφσκι. Μετά θα δώσω το λόγο στους και ηγητές και στη συνέχεια στους υπολείπους βουλευτές. Στο τέλος της συζήτησης θα περιμένω την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε πραγματικά να ξέρουμε πού το πάτε. Θυμίζω την προθεσμία κατάθεσης των τροπολογιών 18 Ιουλίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστώ την προσοχή σας ότι είναι δύο τα είδη των τροπολογιών που μπορούμε να καταθέσουμε. Τροπολογίες στο σχέδιο γνωμοδότησης και τις γνωστές ε, τροπολογίες του προπολογισμού. Για τις ε, προπαρασκευαστικέ δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα υπάρχουν ειδικά έντυπα που θα πρέπει να διαβιβάσετε στη γραμματεία. Όλα αυτά θα ψηφιστούν στη συνεδρίαση της Επιτροπή μα στι 31 Αυγούστου. Λοιπόν, κύριε Σιγητά μου, έχετε το λόγο. Děkuji paní předsedající za udělení slova. Eh, Jsem přihledl k naší minulé debatě s panem Murásem, zpravodajem v pro rozpočet a snažil jsem se... No translation? Δεν υπάρχει διερμηνία. Λοιπόν, είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα χωρίς διερμηνία. Τώρα λειτουργεί η διερμηνία. Τώρα, ναι, εντάξει, ναι, ναι function. Nous avons, vous pouvez reprendre. Excusez-nous, Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Once more, yeah. Επαναλαμβάνω. I minulé debatě s panem Murasanem, zpravodajem v hlavním výboru pro Naonasi. Τι πατάνε οι Άγγλοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό με τη διερμηνία μάλλον. Monsieur Telinska, C'est notre Τελευταία συνεδρίαση είναι. Λοιπόν, οι δερμηνείς είναι εντάξει. Τώρα ακούτε τα αγγλικά, μάλιστα. Τώρα είναι εντάξει, μάλιστα. Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, μια εμπλοκή εδώ. Λοιπόν, ο εισηγητής, ξαναρχίζω. Για τρίτη φορά. Και τρίτη, τρίτη και τυχερή ελπίζω. Όταν ε, συνέτασα τη ε, γνωμοδότησή μου, ε, προσπάθησα να λάβω υπόψη και την προηγούμενη συζήτηση. Συζήτηση που είχαμε κάνει με τον κύριο Μουρεσάν ε, της Επιτροπής των Προϋπολογισμών, ο οποίος είναι ε, αρμόδιος εισηγητής για τον προϋπολογισμό φέτος. Και επίσης ε, προσπάθησα να λάβω υπόψη μου και τα όσα είχαν πει οι συνάδελφοι. Ποια ήταν τα βασικά θέματα που με ενδιαφέραν. Πρώτον, η διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη Connect Europe Facility είναι ένα από τα αγκάθια στη χρηματοδότηση των μεταφορών και καλό ε, είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει σωστή ε, πρικοδότηση και να μην επαναληφθεί η κατάσταση που είδαμε στο παρελθόν ότι παίρνουν τα κονδύλια από το ΣΕΦ για να τα πάνε στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης, ορισμένα έργα χρειάζονται επιδοτήσεις, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση. Και θα πρέπει επαναλαμβανειλημμένα να μιλάμε για τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, ε, χωρίς να λησμονούμε ε, τη σημαντική ε, συνεισφορά των ιδιωτών, ιδιαίτερα στις μεταφορές. Ε, τρίτο, θέμα. Μεταξύ άλλων ε, προτεραιοτήτων, υποστήριξη των διασυνδέσεων μεταξύ των ε, διαφόρων ε, έργων στα ευρωπαϊκά δίκτυα και ιδιαίτερα τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Είμαι πεπισμένος επίσης για τη σημασία του ευρωπαϊκού συστήματος πλοήγησης Γαλιλαίο και Έγνος. Εδώ μπαίνουν και ζητήματα ασφάλειας, ενεργητικής και παθητικής. Εξεπλάγει και εγώ όπως και πολλοί από εσά ε, γιατί προβλέπεται μείωση στο προπολογισμό σε σχέση με την περυσινή πρόβλεψη της τάξης του 9,6%. Στις δημοσιονομικές προοπτικές διαφέρει η χρηματοδότηση από χρόνο σε χρόνο για διάφορους λόγους και αυτό το καταλαβαίνω γιατί όσο προχωρούν τα έργα μπορεί να αλλάζει η χρηματοδότηση αλλά θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί στην χρηματοδότηση τέτοιων έργων όταν τα έχουμε επιλέξει γιατί έχουν αποδείξει την ευρωπαϊκή τους προστιθέμενη αξία. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση για να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Και το ίδιο ισχύει και για τον οργανισμό GSI. Θα συζητήσαμε αυτά την περαισμένα φορά. Ε, τελευταίο θέμα, πέμπτο στη σειρά. Είχα την ευκαιρία να δω το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση για τα πιλωτικά προγράμματα και είμαι πεπισμένος ότι... Μπορούμε να βρούμε κάποια ε, πιλωτικά έργα που στο μέλλον θα γίνουν ε, ουσιαστικά και σημαντικά. Είμαι στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Τώρα το λόγο έχουν οι σκιώδεις. Οι Σιγητές, πρώτος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριος Μαρινέσκου. Uh, opinia prezentată cred că include foarte multe dintre aspectele pe care Comisia Tran ar trebui să le susțină în bugetul pe 2000. Uh. Ευχαριστώ τον εισηγητή και ευχαριστώ και τον κύριο μου. Ε, ε, ε, ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί πιστεύω ότι πολλά από αυτά που είπαμε τα έχει συμπεριλάβει στην, στο σχέδιο γνωμοδότησης. Ως προς το δίκτυο TNT-T ε, και το σκέλος για τις μεταφορές, θα πρέπει να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει σωστός συντονισμός. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται και υποβάλλονται τα σχέδια για κάθε κράτος μέλος. Να γίνει συντονισμός μεταξύ των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής για τους αυτοκινητόδρομους που συνδέουν τα κράτη-μέλη. Εάν τα έργα εντός ενός κράτους συμπίπτουν με τα έργα άλλου κράτους σε ό,τι έχει να κάνει με τη διασυνοριακή πτυχή των θεμάτων αυτών, τότε ε, θα πρέπει να, γίνει, να γίνουν τα κατάλληλα βήματα. Αυτό δεν ισχύει για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Εμείς επιμένουμε. Το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να αξιοποιηθεί για το core και όχι για το comprehensive. Τώρα το, ο Γαλιλαίος είναι άλλο θέμα και πρέπει να το στηρίξουμε. Αλλά και η υπηρεσία της Πράγας πρέπει να υποστηριχθεί από τη στιγμή που το έργο για τον Γαλιλαίο μπαίνει στην τελική του φάση πριν τεθεί ε, σε λειτουργείο. Και η υπηρεσία στην Πράγα χρειάζεται 23 θέσεις απασχόλησης και από αυτές τις 23 θέσεις απασχόλησης έχουν καλυφθεί μόνο οι 5. Ως προς το σύστημα έγνος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα να ζητήσουμε κονδύλια και για την Ουκρανία και για τις χώρες της Βορείου Αφρικής, έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο της επικράτειας της Ένωσης. Καλό θα ήταν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την κατάσταση έτσι όπως, έτσι όπως έχει με τα κονδύλια που χρησιμεύουν για τις στρατηγικές για το Νούμπιο, που θα πρέπει να το εντοπίζει κανείς σε όλη του τη διαδρομή, άρα σε όλη την τροχιά. Άρα να το εργαλείο αυτό να έχει τα κονδύλια που αποφασίστηκαν στην αρχή του έργου. όλα τα κονδύλια του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων να ε, επανεσωματωθούν σε αυτό το εργαλείο για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χάρτσοκ. Τούγκ. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ. Καταρχά, ζητώ συγγνώμη εξ τη κυρία Κραπίνη, που είναι η δική μα εισηγήτρια από Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Οπότε την αντικαθιστώ εγώ. Και θα προσπαθήσω να σα εξηγήσω τη θέση των Σοσιαλιστών. Καταρχά, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για ε, το έργο του, για το σχέδιο γνωμοδότησης, για το σχέδιο Γενικού Προπολογισμού του 2018. Εξ ονόματος της ομάδας μας θα θέλαμε να τονίσουμε ορισμένε προτεραιότητες, οι οποίες επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στις τροπολογίες μας και θα το κάνουμε. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι ο προπολογισμό ε, που δίνεται στις μεταφορές ε, και ε, το τουρισμό θα πρέπει να συνάδει με την ανάπτυξη ε, της απασχόλησης και της οικονομίας στους κλάδους αυτούς. Θα πρέπει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ασφάλεια στις μεταφορές επιβατών σε όλους τους κλάδους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ αντιμετωπίζουν προβλήματα για να προσαρμοστούν στη ψηφιακή αλλαγή και χρειάζονται υποστήριξη. Επίσης, έργα που έχουν να κάνουν με την καινοτομία και την ε, αυτόνομη οδήγηση επίσης πρέπει να υποστηριχθούν. Για τις υποδομές και τις συνοριακές και αυτές είναι για μας ε, προτεραιότητα για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών στην οποία βασίζεται η ιστορική αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθούν κονδύλια έτσι ώστε να ε, διατηρηθεί η υποδομή και να υπακούει σε κάποια κριτήρια και πρότυπα για την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλειά τους. Και εμείς θα κάνουμε προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις για την προώθηση του ε, τουρισμού ε, και των αυτόνομων μεταφορών και την αυτονομία διοίκηση. Προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία με τον εισηγητή. Κύριε Στέλιτσκα. Uh, uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, οφείλω να πω ότι όλοι οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή θα μπορούσα να προσυπογράψω 100% σχεδόν το περιεχόμενο του σχεδίου γνωμοδότησης. Είναι καλά ισορροπημένο, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη του το γεγονός ότι το 2018 είναι κατά πάσα πιθανότητα και η τελευταία ολόκληρη χρονιά κατά τη διάρκεια της θητείας μας, η τελευταία χρήση δηλαδή. Άρα σημαντικό είναι να εστιάσουμε στις δράσεις που θα κομίσουν θέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νομίζω ότι ο εισηγητής το επιτυχάνει. Εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι έχουμε αυξανόμενο προϋπολογισμό για το ESA, για το CESAR και για τα λοιπά. Έχει διατηρηθεί η κατάσταση στο ΣΕΒ και γίνονται τα δέοντα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στο Γαλιλαίο. Δεν θέλω να επαναλάβω τα είδη λεχθέντα. Νομίζω ότι έτσι έχουμε συνέπεια και σωστή ιεράρχηση με αυτά που έχουν προβλεφθεί. Θα περιοριστώ λοιπόν κυρία Πρόεδρε μόνο σε ένα ερώτημα που έχω να απευθύνω. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Γιατί η πρόταση για το προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Συντεροδρομική Υπηρεσία είναι ε, μειωμένη, γιατί ο προπολισμό είναι μειωμένο στην πρόταση. Πώς αυτό συνάδει με τις ανάγκες και πώς αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι έχουμε τότε την τέταρτη δέσμη μέτρων για τις υδροδρομικές μεταφορές, το τέταρτο πακέτο. Σταματώ κάπου εδώ, ζητώ συγγνώμη γιατί δεν θα είμαι σε θέση να ακούσω την απάντηση. Οι συνάδελφοι όμως θα την, ακούσει, θα την ακούσουν και θα μου τη μεταφέρουν. Οφείλω να αποχωρήσω γιατί είμαι συγγητή σε ε, άλλη έκθεση που συζητείται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Ήτρε και σα ζητώ συγγνώμη γιατί θα αποχωρήσω. Ευχαριστώ. Κύριος Κράμε, κατ' εξαίρεση δέχομαι ότι φεύγετε, κατ' εξαίρεση έτσι να φύγετε στο καλό να πάτε και θα περιμένετε και να ακούσω την απάντηση. Εγώ εκπροσωπώ τον Μπάσεκ Χαουτ, τον δικό μας σκιώδη που κολλείται σήμερα και απουσιάζει. Ευχαριστεί και εκείνος και για την έκθεση και για τη συνεργασία. Τρίνε τα θέματα που θέλουν να τονίσουν οι πράσινοι πρώτον τα διασυνοριακά τμήματα που τώρα έχουν γνωρίσει μεγάλη άνθηση. 110 εκατομμύρια επιπλέον βρέθηκαν για τα διασυνοριακά ε, που καταστράφηκαν ε, υποδομές στον πόλεμο και μεταπολεμικά. Εκεί είναι πραγματικά η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Γιατί τα κράτη-μέλη παίρνουν συχνά ευρωπαϊκά χρήματα, όχι ευρωπαϊκά έργα, αλλά για τα εθνικά τους έργα. Δεύτερον, τα νυχτερινά τρένα Τώρα στη Γερμανία καταργήθηκαν πολλά και στο παρελθόν γιατί αυξάνεται το κόστος ε, του δρομολογίου και δεν αποδίδουν τα τρένα, άρα τα καταργούν. Αν το κάναμε αυτό στα αεροπλάνα στην Ευρώπη θα είχαμε ε, το, την ε, κατάσταση ότι θα έκλαιναν τα μισά αεροδρόμια, γιατί τα μισά αεροδρόμια στην Ευρώπη είναι ελληματικά. Άρα θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια για όλους και στα περιφερειακά αεροδρόμια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι μπορούν να έχουν ελλείμματα 10 χρόνια. Στο 11ο ε, έτος κλείνουν. Παρακαλώ να εφαρμοστεί το ίδιο και για τα νυχτερινά τρένα για να μην καταργούνται. Και ε, το τρίτο βεβαίω είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή. Εκεί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο κλάδος των μεταφορών γιατί είναι ο μόνος ε, που δεν έχουν μειωθεί ε, οι εκπομπές από το 1990 παρά έχουν αυξηθεί κατά 22 παρακαλώ Προς τα εκεί θα κάνουμε εμεί τροπολογίε, Γενικά συμφωνούμε όλοι αλλά θα αποκρισταλωθεί και στις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Όλα αυτά εξ ονόματος του Μπάσεκ Χάουτετ. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Κυρία Κονέτσνα, εσάς έπρεπε πρώτα να ακούσουμε. Ζητώ συγγνώμη. Πρώτα εγώ και μετά η πράσινη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Τωσενόφσκι για αυτό το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Εξετάζουμε τις τροπολογίες. Θα ήθελα όμως ε, καταρχάς να αναφέρω κάποιες βασικές παρατηρήσεις που έχω να κάνω και χαίρομαι διότι έχει ασκηθεί ε, επίκριση, κριτική στις περικοπές του ΤΕΝΤΗ είναι ένα πολύ σημαντικό ε, εργαλείο για τη βέλτιστη αξιοποίηση του όλου δικτύου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υφιστάμενες υποδομές θα διατηρηθούν αξιοποιώντας αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και θα βελτιωθούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθούν όλες οι διασυνδέσεις και οι υποδομές που χρησιμεύουν στην διασύνδεση της Ευρώπης. Θα ήθελα να δοθεί περισσότερη προσοχή στο σύστημα Γαλιλαίου και στο έγνος, και από πλευράς ασφάλειας στις αεροπορικές, θαλάσσιες, ναυτιλιακές, οδικές και συνδροδρομικές μεταφορές. Και ο κύριος Στοσινόφσκι και εγώ είμαστε πεπισμένοι ότι είναι απαραίτητη η αποτελεσματική χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Οι περικοπές κατά 7,6% είναι κάτι το εξαιρετικά θλιβερό και λυπηρό. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα εδώ. Και σίγουρα αυτή η νέα πρωτοβουλία για το ίντερνετ δεν θα πρέπει να απειλήσει την ε, συγκρότηση του προϋπολογισμού. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να έχουμε ασφαλείς υδροδρομικές μεταφορές στην Ευρώπη. Οι νέοι θέλουν καταρχάς να επισκεφθούν την Ευρώπη και να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, αυτό είναι σίγουρο, και δεν θέλουν να παγιδευτούν σε ε, συμβάσεις που τους, φέρουν, τους θέτουν σε μειονεκτική θέση. Δεν θα πρέπει το ΕΛΚ λοιπόν να ε, ποντάρει πάνω σε πράγματα που δεν έχουν μια πραγματική αξία και που ουσιαστικά γίνονται σε βάρος της ανάπτυξης. Χαίρομαι για το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Τοσενόφσκη και ελπίζω ότι τα περισσότερα ζητήματα που αντιμετωπίζετε εδώ θα τύχουν στήριξης από την Επιτροπή Μεταφορών και ότι θα είμαστε σε θέση να δείξουμε ότι κάποια πράγματα δεν θα τα δεχτούμε. Περικοπές στη χρηματοδότησή τους. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω τη χαρά εξ ονόματος της Επιτροπής μας να υποδεχθώ και να καλωσορίσω μια ομάδα 17 επισκεπτών, φοιτητών, μαθητών, τους οποίους προσκάλεσε ο κύριος Μικαήλ Καλέ και σας εύχομαι καλώς ορίσατε. Είστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Μεταφορών. Μιλούμε για τις μελλοντικές σας μεταφορές. Επομένως, ε, προσέχετε τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Είστε ευπρόσδεκτοι. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Ρικέ, πυλώνα της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έλαβα την έκθεση από τον κύριο Τουσενόφσκι και τη διάβασα και συμφωνώ σε γενικές γραμμές με το περιεχόμενό του. Καλώς υπογράμμισε τη σημασία των μεγάλων θεμάτων, τη σημασία που έχουν οι επενδύσεις ε, για να βρεθεί αυτή η ισορροπία η δύσκολη μεταξύ των περιφερειακών πολιτικών και των σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων και των πολιτικών μεταφορών και των σχετικών της εργαλείων χρηματοδότησης. Όμως αυτή είναι μία έκθεση για θέματα προϋπολογισμού που θα εξετάσει η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Και υπ' αυτή την έννοια έχω να κάνω κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Αυτό το σχέδιο δηλαδή θα το υποβάλουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να αναφέρθω στο σχόλιο για τη διαστημική πολιτική, για το Γαλιλαίο και το έγνος. Όμως αυτές οι πολιτικές από πλευράς προϋπολογισμού δεν εξαρτώνται από εμάς και από την αποστολή μας. Άρα να το συζητήσουμε, θα ασχοληθούμε με όλα τα σήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό ή μόνο με το σκέλος των μεταφορών στον προϋπολογισμό. Εγώ νομίζω ότι έχουμε αρκετά να υπερασπιστούμε από πλευράς μεταφορών. Σίγουρα συμφωνώ με τη διαστημική πολιτική και την πολιτική για τους δορυφόρους είναι πολύ ενδιαφέρουσε πολιτικέ, αλλά από πλευρά προπολογισμού ή δεν εξαρτώνται από την Επιτροπή μα, την Επιτροπή των Μεταφορών δηλαδή. Και δεν γίνεται και λόγος για τις διάφορες υπηρεσίες και λυπούμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητά μας και μάλιστα αυστηρή. Θεωρώ ότι παίρνουμε πάρα πολύ χρόνο διαβουλευόμενοι για τους κανονισμούς, για τις εφαρμογές τους με τους φορείς που θα τις εφαρμόσουν που είναι οι υπηρεσίες και σε τακτά χρονικά διαστήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της απευθύνω το ερώτημα όπως και οι προηγούμενοι θέλει να αυξήσει τη δουλειά ε, των υπηρεσιών, το φόρτο εργασιών μειώνοντας του ανθρωπίνους πόρου των υπηρεσιών που τις τελεχώνουν και αυτό με προβληματίζει. Είναι σαφέ ότι η δουλειά για την ε, τέταρτη δέσμη μέτρων για τα σιδηροδρομικά έχει ξεκινήσει. Μειώνουμε του πόρου αυτή τη υπηρεσία πώς θα καταφέρει να φέρει αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει και για άλλες υπηρεσίες, για την διαστημική υπηρεσία, όπου μοιράζονται οι πόροι και θα πρέπει αυτό το μοίρασμα να επανεξεταστεί, γιατί κατά κύριο λόγο είναι εξωτερικοί πόροι. Θα μπορούσε, να, θα να εξεταστεί και η παρέμβαση που γίνεται στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να είναι ανάλογο με τη δυνατότητα που έχει να παρεμβαίνει επί τόπου. Εν συντομία λοιπόν, λοιπόν ούτε στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία είναι καλά τα πράγματα, είναι προβλήματα αυτά και πρέπει να επιληφθούν οι αρμόδιοι. Από εκεί και πέρα μου αρέσει πάρα πολύ το σχέδιο Interrail, το λατρεύω και πολλοί από εσά το θεωρούν εξαιρετικό και θαυμάσιο και εγώ το πιστεύω ότι το ακούν και οι, οι φοιτητέ που παρίστανται στην Επιτροπή μας αλλά δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Εγώ δεν το στηρίζω από πλευράς προϋπολογισμού. Είναι ένα project με προϋπολογισμό 3 δις ευρώ, ε, δεν χρηματοδοτείται και υπενθυμίζω ότι το Interrail είναι τριπλάσιο από αυτό που δίδεται ετησίως για το σύνολο της έρευνας και της ανάπτυξης σε θέματα μεταφορών. Μπορεί κανείς να είναι γενναιόδωρος με το Ιντερέλ, το οποίο είναι πολύ συμφέρον και απανηρό για τους ε, φοιτητές. Θα πρέπει όμως ως Επιτροπή να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, γιατί θα έχει αντίκτυπο στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσής μας και θα έχει αντίκτυπο και πιο συγκεκριμένα στον προπολογισμό για τις μεταφορές. Να είμαστε λογικοί και ως εκ τούτου, παρόλο που είναι μια καταπληκτική ιδέα, δεν στηρίζω αυτή την πολιτική από πλευράς επιλογών προπολογισμού. Όμως, για την έρευνα, για την ανάπτυξη πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι να προσδιορίσουμε τα 6,4 δις που αφιερώνονται βάσει ορίζοντα 2020 στις μεταφορές. Αξίζει αυτό να το συζητήσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να συμμετάσχει και να ε, εκφράσει την απόψή της για το θέμα αυτό. Συμμερίζομαι λοιπόν όσα λέει ο εισηγητής με την επιφύλαξη της, ε, του Interrail, ωστόσο να επανέλθουμε στα θέματα του προϋπολογισμού που άπτονται των μεταφορών αποκλειστικά και μόνο. Αυτό περιμένει από εμάς η Επιτροπή Προϋπολογισμού και αυτό πρέπει να κάνουμε. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα υποβάλω επιπρόσθετες τροπολογίες που θα συμπληρώσουν την εξαιρετική δουλειά του κυρίου Τόσονεύσκη. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρόσκληση στη συναδέλφου κυρία Ρούντου Βελών, ε, θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τους εκπροσώπους των οδικών μεταφορών της Εθνικής Ομοσπονδίας Οδικών Μεταφορέων. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας, κυρίες και κύριοι. Η θέση σας είναι εδώ και εδώ για να ακούσετε διάφορα Και εμείς μάθαμε πολλά για το θέμα της οδικής ασφάλειας μετά την ε, έκθεση του μέλους μας. Με μεγάλη χαρά σας βλέπουμε στην Επιτροπή μας. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Στρέφομαι προς τον κύριο Φίλιπ Ρόμπερτς για να ακούσουμε το σύνολο των απαντήσεων. Φίλιπ Ρόμπερτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάρκ Παράν λέγομαι και εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές. Χαίρομαι γιατί υπάρχει αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητή που πηγαίνει προς την κατεύθυνση ε, που επιθυμεί και προσπαθεί να στηρίξει και να ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε δύο-τρία ερωτήματα που μου έχουν τεθεί. Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι η τρίτη πρόσκληση υποβολής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρουσιαστεί αύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή Μεταφορών. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν αύριο και ελπίζω πραγματικά να πάνε προς την κατεύθυνση που ε, παρουσίασαν οι διάφοροι παρεμβαίνοντες που πήραν το λόγο. Να σας πω ότι σε επίπεδο υπηρεσιών που είναι πράγματι τα εργαλεία και οι οντότητες που είναι εξαιρετικά σημαντικές και χρήσιμες για την εφαρμογή της πολιτικής μας, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής εργασίας για την εφαρμογή του προϋπολογισμού κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση για τις εκάστοτε και επιτόπου και επιμέρους ε, λεπτομερείς ανάγκες της κάθε υπηρεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε όλα τα διοικητικά συμβούλια, σε όλες τις προπαρασκευαστικές επιτροπές που συνέρχονται και συνεδριάζουν. Προφανώς δεν μπορούμε να καλύψουμε πάντοτε όλες τις ανάγκες που μας υποβάλλονται και που μας ζητούνται, αλλά πλησιάζουμε πολύ. Είμαστε πολύ κοντά. Και πρέπει να τηρήσουμε και τα δέοντα σε σχέση με τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Επομένως, οι ανάγκες που ταυτοποιήθηκαν και αναγνωρίστηκαν για το 2018 ε, φαίνεται ότι οι πόροι που διατίθενται θα είναι επαρκείς. Βεβαίως είμαστε πάντοτε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι προς το παρόν δύσκολο και γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά φαίνεται ότι οι πόροι είναι επαρκείς για να ε, φέρουν σε πέραση ε, αρμόδιοι τα καθήκοντα που ε, έχουν αναλάβει. Επομένως με θετικό βλέμμα, με θετική ματιά πρέπει να τα βλέπουμε αυτά και σίγουρα πάντοτε κανείς χρειάζεται περισσότερους πόρους, ποτέ δεν θα περισσέψει κανείς πόρους. αυτό είναι βέβαιο. Από εκεί και πέρα για τα πιλωτικά προγράμματα έχουμε το παράρτημα 4 στον προϋπολογισμό, το οποίο παρουσιάζεται αποτελέσματα. Αν έχετε όμως συγκεκριμένες ερωτήσεις για κάποιο φάκελο συγκεκριμένο, είμαστε στη διάθεσή σας για να προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Ρόμπερτς, μας είπατε ότι αύριο θα μας παρουσιάσετε τα αποτελέσματα. Όμως θα μας παρουσιάσετε τα αποτελέσματα για το μηχανισμό διασύνδεσης. Για τα άλλα θέματα μπορούμε να έχουμε θέση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν συντομία, μια κάποια θέση να μάθουμε τη δική σας. Και επίσημη θέση της Επιτροπής, που θα βοηθήσει τον εισηγητή μας. Υπάρχει προθεσμία, υπάρχει χρονοδιάγραμμα. I wasn't expecting to speak. Ε, Δεν περίμενα πάρα το λόγο. Αύριο θα σας ε, παρουσιάσουμε τη μελέτη, θα το συζητήσω με τον διευθυντή μου και αύριο θα σας φέρουμε τις λεπτομέρειες, αν συμφωνείτε. Μάλιστα. Όλοι ακούσατε ότι αύριο θα έχουμε μία λεπτομέρεια σε σχέση με τους οργανισμούς. Ευχαριστώ, Κομισιόν. Ας ξαναδώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως όλους τους συναδέλφους τις εισηγητές για τα καλά τους λόγια. Μία επιπλέον πληροφορία Κατανοούμε ότι είναι πολύ σημαντική η σύνδεση ανάμεσα στους οργανισμούς ε, GSA και έγνος ε, για το μέλλον. Για παράδειγμα, για το σύστημα διοδίων η δυνατότητα χρήσης ε, του συστήματος ΙΤΟ είναι πολύ σημαντική. Αυτό το είχα τονίσει και στην έκθεσή μου. Τώρα υπάρχει, γίνεται μάλλον μια παρόμοια συζήτηση και στην Ήτρε για το προϋπολογισμό ώστε να φανεί ότι είναι πραγματικά αλληλένδετα αυτά τα προγράμματα. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, ώστε να μπορέσουμε όλα αυτά να τα εντάξουμε στο κείμενο και να βελτιώσουμε την ε, ε, έκθεση. Ελπίζω λοιπόν πως θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτική αυτή η έκθεση για την Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τοζενόφσκι για κατάθεση τροπολογιών. Έχουμε προθεσμία 18 Ιουλίου το μεσημέρι. Συνεχίζουμε τώρα τις εργασίες μας με την έκθεση για τη διάσωση ζώων και αύξηση της ασφάλειας των αυτοκινήτων σε συνεργασία με την ΕΜΚΟ. Ο, ο εισηγητής μας είναι ο κ. Κοχ. Θα του δώσω το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στους Κιώδης και θα ζητήσω και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Κοχ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Το ξέρουμε εδώ και καιρό. Η οδική ασφάλεια εξαρτάται από τρεις παράγοντε. Πρώτον το όχημα, Δεύτερον, τι υποδομές και τρίτον ε, τη συμπεριφορά του οδηγού. Άρα χρειάζονται μέτρα και στους τρεις τομείς για να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια. Ακόμα και αν αυτό που μας απασχολεί σήμερα στο πλαίσιο της έκθεσης είναι η ασφάλεια του οχήματος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να μιλήσουμε για γενικότερες απαιτήσεις για την οδική ασφάλεια, γιατί ε, αλληλεπιδρούν όλα αυτά τα μέτρα. Άρα, εγώ θα ήθελα μεγαλύτερο έλεγχο στους αυτοκινητοδρόμους. Μας λένε ότι δεν έχουν υπαλλήλους. Ε, υπάρχουν συστήματα τεχνικής βοήθειας για τους ελεγκτές και Επίσης, μπορεί να γίνει και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και ευφυών τεχνικών. Εδώ γίνεται ήδη πολύ καλή δουλειά, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν πολύ περισσότερο. Γενικά τώρα το σύστημα ε, επικούρησης της οδήγησης. Αυτά τα συστήματα ε, διευκολύνουν ε, την, και αυξάνουν την ασφάλεια την οδική γιατί το 95% των ατυχημάτων και των δυστυχημάτων οφείλονται ε, σε συμπεριφορά του οδηγού ή σε λαθασμένη εκτίμηση. Επίση, μειώνεται η κατανάλωση των καυσίμων ε, ε, και είναι και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που έχουν περιορισμένη κινητικότητα. Γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ρυθμίσεις ε, για να βελτιστοποιηθούν τα συστήματα αυτά, τα αυτόματα συστήματα βοήθειας της οδήγησης. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει ο οδηγός να κατανοεί ε, τα συστήματα που ακούει τα ηχητικά σήματα ε, και να τα αναγνωρίζει. Γιατί πολλές φορές τον εκνευρίζουν όλα αυτά που ε, σφυρίζουν και χτυπάνε και τα κλείνει. Άρα δεν υπάρχει βοήθεια στην οδήγηση. Σε ό,τι αφορά την ειδική βοήθεια και τα ειδικά συστήματα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνο εκείνα τα οποία έχουν τις εξής τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, θα πρέπει να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη η ουσιαστική συνεισφορά του στην αύξηση της οδικής ασφάλειας. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι θετικό το ισοζύγιο κόστους ωφέλειας και τρίτον, θα πρέπει να είναι όριμα για να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα, στα πλαίσια της δικής μου έκθεσης προτείνω εννέα μέτρα ε, ενεργητικής και παθητική ασφάλειας που κατά την άποψή μου θα πρέπει να τα λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που ελπίζω να φέρει την πρόταση για τον αντίστοιχο κανονισμό αρχές του 2018. Δεν θέλω να σας αναφέρω και τα εννέα μέτρα, δύο μόνο. Όποια μέτρα ασφαλείας και να έχουμε θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή ε, στους πιο ασθενείς ε, οδηγούς και μας πιο ηλικιωμένους πολλές φορές που πρέπει να προστατεύουμε και να λαμβάνουμε υπόψη το αυτόματο φρένο ε, ασφαλείας και κινδύνου είναι πολύ σημαντικό διότι μπορεί να μειώσει και να αποφύγει πολλά ε, δυστυχήματα. Βοηθάει λοιπόν αυτό το σύστημα να αξιοποιηθεί πλήρως η ε, δυνατότητα του αυτοκινήτου φαινός και να αποφεύγονται οι απροσεξίε ή αμέλειε των οδηγών. Υπάρχουν ορισμένα συστήματα που είναι υποχρεωτικά, ε, αλλά θα πρέπει να μεταξελιχθούν και να αναπτυχθούν. Αυτά ισχύουν για τα φορτηγά, αλλά για τα χρήσεις χρήσεως και τα ε, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ε, δεν υπάρχουν αυτές οι ρυθμίσεις ε, όπως είναι ε, αυτόματη αναγνώριση πεζό και ποδηλατών. Θα πρέπει λοιπόν και στα γιοταχή και στα φορτηγά και στα λεωφορεία και στα μικρά επαγγελματικά οχήματα. Πολλές φορές οι πολυδηλάτες και οι πεζοί βρίσκονται στην νεκρή γωνία, στην τυφλή γωνία του αυτοκινήτου και δεν τους βλέπουν οι οδηγοί. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάμερες, αισθητήρε ε, και λοιπά ε, συστήματα αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών και ε, στα γιοταχή και στα φορτηγά και στα λεωφορεία. Συνειδητά δεν ανέφερα προθεσμίες μέχρι πότε θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ποια συστήματα που βοήθησης της Αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Ε, η έκθεση μου είναι έκθεση πρωτοβουλίας και θα πρέπει κυρίω να αφοσιωθεί ε, στα ποια είναι εκείνα τα μέτρα που πρέπει να είναι υποχρεωτικά ενεργητικής και παθητική ασφάλεια και όχι μέχρι πότε θα τα επιβάλλουμε. Θα παρακολουθήσω την προσοχή σας, ε, κυρία Πρόεδρε. Αυτό το τελευταίο θέμα θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να το λύσουμε όταν συζητήσουμε τον κανονισμό γενικής ασφάλειας σε συνεργασία με την Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς. Και τέλος, ένα σύντομο σχόλιο. Ε, στα γερμανικά έχω κάνει το σχέδιο έκθεσης. Στην αγγλική μετάφραση ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλά μεταφραστικά λάθη που αλλοιώνουν το περιεχόμενο και που θέλω να βελτιώσω με κάποιες τροπολογίες. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο σύστημα υποβοήθησης που σταματάει το ίχνος ένεργα ε, και ένα άλλο το, το οποίο ενημερώνει για ε, το ίχνος που αφήνει πίσω του το όχημα. Στα αγγλικά έχει μεταφραστεί λάθος αυτό. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα που δεν χωράνε σε μια έκθεση πρωτοβουλία. Η προθεσμία κατάθεση είναι πολύ μικρή λόγω και των θερινών διακοπών. Λίγη την Παρασκευή τώρα στις 11 η ώρα. Στις 14 του μηνός. Εγκαίρως όμως έστειλα το κείμενο στους συναδέλφους για να μπορέσουν να το μελετήσουν και να ετοιμάσουν τις τροπολογίες τους. Ε, με χαρά περιμένω τα σχόλια και τη συνεργασία με τους ηγητές και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci, Monsieur Koch. Je vais demander à la personne qui... Euh, ε, ζητήσω από όσου ε, συμμετέχουν, βρίσκονται στην αίθουσα, μάλλον να σβήσουν τα τηλέφωνά τους ή να τα βάλουν στη δόνηση. Λοιπόν, να πρέπει να έχουμε πέρα από τα κείμενα και τις δηλώσεις των Υπουργών ε, στην Μάλτα δράση. Γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε νούμερα και κυρίως τον αριθμό των θυμάτων. Δηλαδή 26.000 ε, νεκροί στους δρόμους μας. Δεν το λέμε όμως αρκετά ότι το γεγονός ότι έστω και ένας νεκρός ε, στους δρόμους σημαίνει άλλους 7 ανάπηρους. κόστος για την κοινωνική πρόνοια και κόστος σε ζωές. και σε τραυματίες. Γι' αυτό Γι' αυτό και πρέπει να τονίσουμε αυτό το ζήτημα τώρα. Πρέπει δηλαδή να περάσουμε στη δράση. Αυτό ήθελα εγώ να πω για να στηρίξω αυτή την έκθεση. Και δίνω το λόγο στην κυρία Σινιάλοβα. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Ε, δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτή την έκθεση. Αμα, πέρα όμως από τα μέτρα για τη βελτίωση το, της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές και την επιβολή καλύτερης συμπεριφοράς στους οδηγούς, θα πρέπει να μιλήσουμε και για το κοινωνικό πλαίσιο, όπου πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά το θέμα της ασφάλειας, ώστε... Ε, να μπορέσουμε να, μιλώσουμε, να μειώσουμε στο μηδέν τον αριθμό των νεκρών. Συμφωνώ με για το γεγονός ότι η Κομισιόν θα πρέπει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να υποβάλει ε, έκθεση για τη γενική ασφάλεια και για την οδική ασφάλεια και Πιστεύω ότι θα πρέπει να υποβάλουμε και μια τροπολογία για την προστασία των πεζών, γιατί είναι η πιο ευάλωτη. Πρέπει να προστατεύονται. Και τα συστήματα βοήθεια των αυτοκινήτων, οι ειδοποίησει θα πρέπει να εστιάζουν την προσοχή στους πεζούς για να μειωθούν τα ατυχήματα. Επίση, οι δοκιμές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ε, θέση των ε, πεζών ε, θα πρέπει επίσης τα συστήματα έγκυρης ειδοποίησης να δοκιμάζονται. Συμφωνώ και σε αυτό με τον εισηγητή. Το κείμενο του είναι πολύ ισορροπημένο και περιλαμβάνει τις προτεραιότητές μας και όπως και στο παρελθόν προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους σκιώδες εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Merci, Madame la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 θέλω να όντω συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει από κοινωνική και οικονομική άποψη να μεριμνήσουμε. Γι' αυτό και συμφωνώ με τον εισηγητή για τα αιτήματά του ε, να υπάρξουν στοιχεία όσον αφορά τους ποδηλάτες, ε, τους ηλικιωμένους και τους πεζούς. Έχουν γίνει πολλά πολλά ε, όσον αφορά τα ίδια τα αυτοκίνητα για να βελτιωθεί η ασφάλεια των πεζών και των ποδηλατών, αλλά πρέπει να ε, ασχοληθούμε και με τις νεκρές γωνίες του αυτοκινήτου αλλά και με τα ατυχήματα που οδηγούν σε μόνιμη αναπηρία. Ιδιαίτερα τα φορτηγά είναι υπέτεια τακτικά για μεγάλα προβλήματα, μεγάλα ατυχήματα και κυρίω όταν κυκλοφορούν εντό των πόλεων. Από αυτή την άποψη πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τη τεχνολογία, όσο και προηγμένη να είναι, και να ειδοποιεί τον οδηγό δεν ε, ε, καλύπτει τα πάντα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται διάφορες συσκευές που επιτρέπουν στον οδηγό να βλέπει καλύτερα το δρόμο, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά αυτοκίνητα είναι παλιά. Και αυτά τα παλιά αυτοκίνητα προκαλούν πολλά ατυχήματα και θύματα σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Πολωνία. Και θα πρέπει να δούμε πώ θα βελτιωθεί η ασφάλεια και για αυτά τα αυτοκίνητα, προωθώντα τι σωστέ τεχνολογίε που επιτρέπουν στον οδηγό να μπορεί να αντιδράσει πιο γρήγορα και με ένα παλιό αυτοκίνητο φυσικά. Προβλέπουμε, προβλέπουμε στο μέλλον με προδιαγραφές ε, για τα επόμενα 3-5 χρόνια, αλλά πρέπει να δούμε και το παρόν. Μπορεί να κοστίζει, αλλά σίγουρα είναι απαραίτητο. Εκτός από αυτά λοιπόν δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν προβλέπουμε να υποβάλουμε πολλές τροπολογίε. Είμαι ευτυχής που θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και με τους υπόλοιπους σκιώδεις για αυτήν την τόσο σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζερικέ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι εξαιρετική έκθεση. Πρέπει αυτό να το πω εξ αρχής. και θέλω να κάνω μόνο κάποιες παρατηρήσεις και να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Το πρόβλημα της ε, ενσωμάτωσης ορισμένων ε, συσκευών στο όχημα ε, είναι θέμα κόστους. Χρειάστηκαν 25 χρόνια ώστε να καταστεί υποχρεωτικό το σύστημα φρένου ABS στα αυτοκίνητα. μάλλον πίσω από αυτό το σημείο δυσκολευόμαστε να δεχτούμε ότι το θέμα της ασφάλειας σε ένα αυτοκίνητο εξαρτάται από το αν μπορείτε να το πληρώσετε. Υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί. Δηλαδή οι φτωχοί ε, ας κυκλοφορούν ε, ε, κινδυνεύοντας, ενώ οι πλούσιοι όχι. Υπάρχει ένα προβληματάκι λοιπόν για το ποιε θα πρέπει να είναι οι συσκευές, όπου θα πρέπει να γίνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να γενικευτεί η χρήση τους, να γίνουν προσπάθειες για μείωση του κόστους τους κτλ. Γιατί όταν μιλάμε ας πούμε, για επιδοτήσεις των κρατών μελών για οχήματα που έχουν μικρότερο αποτύπωμα σε άνθρακα, σωστό και σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να το συζητήσουμε και για τέτοιες συσκευές, ε, μηχανισμούς που έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία. ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ισότητα στα ατυχήματα. Γιατί με ενοχλεί το ότι ξέρω ότι αν κανείς οδηγεί μια μεγάλη Mercedes είναι ασφαλής, ενώ όταν οδηγεί ένα μικρό φιατάκι κινδυνεύει. Είναι η πραγματικότητα αυτή, κοστίζουν ακριβά όλα αυτές, όλες αυτές οι συσκευέ, αλλά πάντως πρέπει να το συζητήσουμε. Άλλη παρατήρηση, πιστεύω ότι πρέπει επίσης να επιμείνουμε για την ευθύνη των υποδομών. Υπάρχουν κάποια μέρη και ε, ανάλογα με το ποιος είναι υπεύθυνο, περιφέρεια, η πόλη, το κράτος, Υπάρχουν ε, μέρη που είναι εγκαταλελειμμένα, υπάρχει ε, πρόβλημα και έχει τονιστεί, το έχουμε πει. Και το λύνονται βάζοντας ακόμα μια πιναγίδα που λέει προσοχή, προσοχή. Ε, υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι απαράδεκτες για το πω και ήπια. Λοιπόν, εφόσον διακρίνουμε ανάμεσα σε έναν δρόμο με δύο λωρίδες και, μια, και ένα αυτοκινητόδρομο, οι πιθανότητες να υπάρξουν ατυχήματα είναι 17 φορές περισσότερος στον δρόμο με τις δύο λωρίδες. Και όταν ξέρουμε πόσο κοστίζουν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί στον προϋπολογισμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών γενικά, ε, νομίζω ότι θα μας αναγκάσει αυτό να κάνουμε κάποιες ε, αλλαγές στις υποδομές εκεί όπου χρειάζεται. Τρίτη παρατήρηση είναι η σήμανση. Εδώ τα κρατημέλη έχουν, φέρουν μεγάλη ευθύνη γιατί που και που η σήμανση είναι ακατανόητη και απλώ προσθέτουν και άλλες πινακίδες, τη μία πάνω από την άλλη και κάθε φορά έχουμε την εντύπωση ότι οδηγεί σε πλήρη αποδιοργάνωση αυτό το πράγμα. Και βλέπω και τον σύντροφο Βίμ Μπαντρικάμ που είναι μοτοσυκλετιστής. Στο Βέλγιο, ας πούμε, εξακολουθούν να μπαίνουν ε, κάποιες φραγμές, κάποιοι φραγμοί κάποιες μπαριέρες που πέφτουν και μπορούν να λειτουργήσουν ως και για τους μοτοσυκλετιστές, θα έπρεπε αυτό να έχει απαγορευτεί τελείως ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι τόσο περίπλοκο. Θα πούμε ότι δεν θα βάλουμε πια άλλο τέτοιο είδους μπαριέρες γιατί ότι Γιατί τα είδα στον ε19, στον ε40. Τώρα, Κάτι ακόμα όσον αφορά την ε, μελέτη των ατυχημάτων. Η διαχείριση της κυκλοφορίας είναι ένας παράγοντας ροής, ε, μείωση των συμφορήσεων και των εκπομπών, αλλά υπάρχει και ο παράγοντας μείωση των ατυχημάτων και η επικοινωνία μεταξύ του οχήματο και της υποδομής είναι πολύ σημαντική. Η, η ενημέρωση για την κατάσταση κυκλοφορίας είναι ένα θέμα καθοριστικό νομίζω. Όπως και οι συσκευές ε, που χρησιμοποιούνται από τα αυτοκίνητα. Πολύ καλά μετρημένη έκθεση αυτή. Δεν έχω να πω τίποτα για τα όσα προτείνονται. Όλα είναι λογικά. Σχεδόν τίποτα δεν έχουμε ξεχάσει. Εγώ υπογράμμισα απλά κάποια στοιχεία που θεωρώ ήταν σημαντικά, αλλά είναι εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κονέτσνα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για το έγγραφο αυτό, γιατί είναι σημαντική και πολύ σοβαρή η δουλειά του. 26.000 άνθρωποι βρίσκουν το θάνατο κάθε χρόνο στους ευρωπαϊκούς δρόμους. 135.000 άνθρωποι ε, τραυματίζονται σοβαρά κατά την οδική τους μεταφορά θα προσπαθήσουμε και θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτά τα νούμερα και να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια. Θα ήθελα η έκθεση να δώσει μεγαλύτερη σημασία στα φορτηγά, τα διαφόρων ειδών φορτηγά, γιατί τα ατυχήματα που, στα οποία εμπλέκονται φορτηγά οδηγούν σε 4.000 θύματα, που και πολύ συχνά είναι ποδηλάτες ή πεζοί τα θύματα. Στα φορτηγά υπάρχουν πάρα πολλές τυφλές γωνίες, οι οδηγοί κάθονται πάνω στη μηχανή και μπορούν να δουν το δρόμο όταν οδηγούν εκτός πόλεων, όμως το ότι είναι πάνω από τη μηχανή και είναι περιψωμένη είναι πολύ επικίνδυνο όταν οδηγούν εντός ε, του άστεως. Τα φορτηγά, για παράδειγμα, στο Λονδίνο συνδέονται με ε, πρόκληση ατυχήματος στα οποία υπήρχαν 35 ποδηλάτες, για παράδειγμα, ε, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν αναγνωρίζονται τα ε, διαφορετικά είδη οχημάτων από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι λυπηρό. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, να πούμε ότι είναι ε, τελείως διαφορετικό ένα μικρό φορτηγάκι, απλό φορτηγό ή ένα ρημολκούμενο όχημα με ρημολκό και ρημολκούμενο αρθρωτό δηλαδή όχημα θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες φορτηγών, βαρέων οχημάτων και να μειωθούν οι τυφλές γωνίες στις οποίες ο οδηγός δεν έχει οπτική πρόσβαση. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να είναι πιο ασφαλείς οι οδικές μεταφορές. Αν ο οδηγός δεν είναι σε θέση να δει τους πεζούς ή τους ποδηλάτες, τότε η θέση τους είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Ε, πρέπει να κάνουμε το παν για να βελτιώσουμε την κατάστασή τους. Ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί μας ευστά την προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Τα έχει περιλάβει στο σχέδιο έκθεσή του και πιστεύω ακραδάντως ότι με του λοιπού και ό,τι συζητητέ θα ε, γίνει το παν για να υπάρξει κατάλληλη μέρημνα για αυτό το ζήτημα. Είναι ένα από του πιο σημαντικού φακέλους για την Επιτροπή Μεταφορών γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια Ευρωπαίων πολιτών, με την ασφάλεια όλων μα τελικά. Γιατί όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το σύστημα μεταφορών. Ο κύριος Κράμερ, ευχαριστώ. Καθυστέρησα λίγο λόγω διαρμηνίας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον εισηγητή, όχι μόνο για αυτά που έγραψε στην έκθεσή του, αλλά και για αυτά που είπε στην αρχή, ότι χρειάζονται περισσότεροι έλεγχοι. Ιδιαίτερα και ο νόμος που δεν ελέγχεται είναι περιττός. Οπότε υπάρχουν ε, διαφορές, θα μου πείτε, μεταξύ κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων πόλεων. Στο Βερολίνο είναι 6-7 οι αρμόδιοι για να κάνουν τους ελέγχους για την ταχύτητα. Στο Βραντεμβόργο το γειτονικό κρατήδιο που έχει ένα εκατομμύριο ε, κατοίκους παραπάνω έχει πενταπλάσιο ξεπλάσιο ρυθμό υπαλλήλων. Μιλήσαμε για τους ασθενείς χρήστες, ε, τους ποδηλάτες, τους πεζούς. Τα ξέρω και εγώ ποδηλάτης είμαι. Στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο ένα ε, λεωφορείο ε, ε, προσπέρασε ένα ποδηλάτι και πάλι λίγο να τον πατήσει αυτός που ερχόταν από την άλλη μεριά. Τα συστήματα έκτακτης πέδησης, τα φρένα αυτά, γιατί είναι καλά, αλλά γιατί έχετε αυτή την πρόταση στη Γερμανία, έγινε ένα φρικτό δυστύχημα της προάλλης στην Νότια Γερμανία και κανονικά μειώνεται η ταχύτητα ε, σε 20-25 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά δεν κοκαλώνει το όχημα. Επίσης, η προειδοποίηση για τις ταχύτητες ε, είναι πολύ καλή, γιατί εκτός από την επίρρεια αλκοόλ, ε, άλλη σημαντική αιτία δυστυχημάτων είναι η υπερβολική ταχύτητα. Ακριβώς επειδή έχει προχωρήσει η τεχνολογία, όταν διαπιστώνεται αυξημένη ταχύτητα, θα πρέπει να έχει ένα κόφτη, να μειώνεται η ταχύτητα. Δεν θα σου ανάβει ένα λαμπάκι ή θα ακούσει ένα κουδουνάκι Παρ' όλα αυτά, θα τρέχουμε 80, 90, 160 όπως έτρεχε ο άλλος προς τις προάλλες πάλι σε μια ζώνη που ήταν 30 χιλιόμετρων την ώρα. Και εκεί θα πρέπει να ισχύει το ίδιο δίκαιο για όλους. Είχα πάει ε, στη Siemens και οδήγησα ένα τρένο υψηλής ταχύτητας με ETMS ε, στο προσωμιοποιητ στα 120 χιλιόμετρα ε, και δεν μπορούσα να πατήσω παραπάνω γιατί ήθελα να στρίψω έτσι με φόρες σε μια ε, απότομη στροφή για να τους δείξω ότι μπορώ να πάω παραπάνω από 120 αλλά δεν μου το επέτρεπε το σύστημα. Γιατί να γίνεται αυτό στη σταθερή τροχιά στο σιδηρόδρομο που είναι πολύ μικρότερη η κίνδυνη ατυχήματος ε, από ότι στον αυτοκινητόδρομο και να μην γίνεται στον αυτοκινητόδρομο. Υπάρχουν πολλά συστήματα πολύ καλά τα έχετε απαριθμίσει όλα, δεν λείπει κανένα και ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά υπάρχει δυνατότητα για τον οδηγό να τα απενεργοποιήσει αυτά τα συστήματα. Μόλις ξέσπασε το, το σκάνδαλο diesel, εκεί υπήρχαν κάποια συστήματα που έπρεπε να φροντίζουν να περιορίζονται οι ρήποι και εκπομπές κτλ. Αλλά τι κάνανε, βγάζανε και καταργούσαν τα συστήματα αυτά. Άρα γιατί να έχω ένα σύστημα προειδοποίησης ή ένα σύστημα πέδησης που να μπορεί να απενεργοποιείται. Για ποιο λόγο να μπορεί κάποιος να το απενεργοποιεί, δεν το καταλαβαίνω. Μετά, για το κόστος. Το είπε και το Κρικέ. Προφανώς. Αλλά έγινε και μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης πριν από κάποια χρόνια ότι κάθε αυτοκίνητο χρηματοδοτείται από το φορολογούμενο στην Ευρώπη κατά 1.600 ευρώ, εάν υπολογίσεις και το παρεπόμενο κόστος. Και εδώ το κόστος ε, ε, είναι και τα δυστυχήματα. Τα πληρώνουν αυτά τα ταμεία, τα ασφαλιστικά, αλλά μέχρι ένα ποσό. Από εκεί και πέρα τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Και αυτά που χρειαζόμαστε είναι ψίχουλα ως κόστος για να βάλουμε τα συστήματα που πρότεινες. Και ένα τελευταίο. Ας πούμε, συζητάμε ε, για τα φορτηγά, για τους καθρέφτες, για να μην υπάρχουν τυφλές γωνίες. Θυμάσαι από πότε, πάνω από 10 χρόνια που είμαστε και δυο εδώ. Και κάποια στιγμή αν δεν μπουν οι πολιτικοί ότι τώρα ε, θα ε, επιβληθεί αυτό, δεν μας παίρνουν στα σοβαρά. Και ξέρουμε πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να σωθούν, πόσες ζωές, ακριβώς και μόνο λόγω αυτής της τυφλής γωνίας στα φορτηγά. Και γενικότερα. Ε, Περιμένω και εγώ την καλή σίγουρα συζήτηση που θα έχουμε για να καταλήξουμε σε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Ο κύριος Φαν Μίλτεμπερχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, του Γιάννη Ρόντε, του σκιώδη ηγετή των φιλελευθέρων που δυστυχώ απουσιάζει, θα ήθελα να πω και εγώ μερικά πράγματα. Και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή. Είναι πάρα πολύ ε, περιστατωμένη η έκθεσή του. Το έχουν πολλοί επαναλάβει ότι έστω και ένα θύμα ε, από τροχαίο είναι ένα θύμα που δεν θα έπρεπε να έχουμε. Από το 2014 δυστυχώς και στη δική μου τη χώρα, στις κάτω χώρες, θρυνούμε πολλά θύματα και αύξηση των νεκρών στην άσφαλτο. Είναι καλά τα μέτρα που προτείνει και συμφωνώ ότι μπορεί με έξυπνο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα πιο αποτελεσματικά ε, μέσα και μέτρα να υιοθετήσουμε. Η οδική ασφάλεια στην Ευρώπη όμως δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το πορτοφόλι ε, του εκάστοτε Ευρωπαίου πολίτη. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συστήματα προειδοποίησης ε, και τα αυτόματα φρένα έχουν μειώσει κατά 5.000 τα θανατηφόρα τροχέα. Ε, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις που σώζουν πραγματικά ζωές. Επίσης όμως έχει σημασία και οι υποδομές οδικές και θα πρέπει εκεί να εστιάσουμε πάρα πολύ. Και υποδομές για πεζούς και ποδηλάτες. Είναι διαφορετικές οι ροές των οχημάτων και έχουν διαφορετικές επιπτώσεις ε, και σε μια χώρα ποδηλατών όπως είναι η Ολλανδία εμεί έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Κοιτάξτε στις Βρυξέλλες, εγώ δεν τολμάω όχι ως ποδηλάτης, ως πεζός να πατήσω το πόδι μου στην άσφαλτο, κινδυνεύει η ζωή μου. Επίσης, και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, είμαι σκιώδης ηγητής για αυτό το θέμα και ε, μας απασχολούν κάποια θέματα. Ε, το επίπεδο φιλοδοξίας θα πρέπει να είναι υψηλό. Ε, θα πρέπει όμως να υπάρχει προστασία των δεδομένων, να υπάρχουν διάφοροι έλεγχοι, τα είπαμε όλα αυτά, και για τις φιλοδοξίες και για τον πύχη. Ε, όταν όσο προχωράει μάλλον η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση ε, των οχημάτων, υπάρχουν και πολλά δεδομένα που μεταδίδονται. Γι' αυτά τα, τα λέει στην παράγραφο 15 ο εισηγητής για τον κανονισμό για τη γενική προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή. Διάβασα στην ανακοίνωση ότι μοιράζουμε διάφορα αστέρια στα οχήματα. Αλλά τουλάχιστον το 1 πέμπτο δεν ανταποκρίνεται στην κατάταξή τους. Υπάρχουν κάποια στοιχεία ασφαλείας που δεν συμπεριλαμβάνουν σε όλα τα αυτοκίνητα. Και η Ευρώπη έχει διαφορετικούς καταναλωτές και διαφορετικές φορολογικές επικράτειες που δεν έχουν όλοι την ίδια αγοραστική δύναμη για να αγοράσει το πιο ασφαλές αυτοκίνητο. Αλλά όταν έχουμε ένα σύστημα απονομής έτσι αστέρων ανάλογα με την ασφάλεια, θα πρέπει αυτό να είναι ασφαλές το ίδιο και ακριβές. Τέλος. Όταν πρόκειται για τα αυτοκίνητα και την κυκλοφορία... Ε, το αλκοόλ, η κατανάλωση νοπνεύματος ε, δεν ε, συνάδει με την οδήγηση. 0% καθόλου αλκοόλ, λέει ο εισηγητή για του επαγγελματίε οδηγού και του νέου οδηγού μέχρι να συμπληρώσουν την πρώτη διετία οδήγηση. Και εναρμόνιση ε, των διαφόρων ε, τιμών ε, που επιτρέπονται ε, να ανοιχνεύονται στι εξτάσεις αίματος. Στα αγγλικά λέγεται αυτό close to zero, αυτό που θέλω να επιτύχουμε, δηλαδή είναι σχεδόν μηδενικό. Και τότε μπορούμε να σηκώσουμε το ποτήρι μας και να κάνουμε μια πρόποση, να πούμε στην υγεία σας. Ο κύριος Βαχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ich ähm, Θα ήθελα να ευχαριστήσω äh, και εγώ τον συνάδελφο Ντίτερ Κοχ για την έκθεσή του και για τις εξηγήσεις του. Ήταν πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και πλήρης η έκθεση. Θέλω να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ζητήσω το εξή. Ε, δείξτε λίγο περισσότερη φιλοδοξία. Το είπε και η πρόεδρο τη Επιτροπή μα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέχρι το 2018 θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτέ τι ε, ε, δράσει. Αλλά ε, λυπάμαι για αυτή την καθυστέρηση. Ε, για την ίδια την έκθεση δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειε για τα διάφορα συστήματα, διότι πρώτον ο δίτερ Κόχ έχει περιγράψει και εξηγήσει όλα αυτά θαυμάσια και επίσης και οι διάφοροι συνάδελφοι είπαν τα σημαντικότερα για τα συστήματα τη οδήγηση για τα συστήματα ασφαλείας και ολόκληρο το πακέτο. Εγώ έτσι το βλέπω ως μια δέσμη ε, μέτρων ασφαλεία και πολλά έχουν ήδη υποθεί. Τώρα, η επικεφαλίδα, ο τίτλος της έκθεσης είναι για μένα κάπως περιορισμένη. Μου το είπε και ο συνάδελφος Βαντενκά. Εδώ τι λέμε. Ενίσχυση της ασφαλείας των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διάσωση ζώων. Αλλά όλοι οι συνάδελφοι και ο ίδιος ο εισηγητής μίλησαν ε, για ένα ευρύ φάσμα μέτρων. Δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των αυτοκινήτων, αλλά ε, και των υποδομών κυρίως, αλλά και την οδηγική συμπεριφορά. Ειδικά οι υποδομές θα πρέπει να μας απασχολήσουν και να μας προβληματίσουν και να είμαστε λίγο πιο προνοητικοί. Γιατί αν κατασκευάζονται σήμερα δρόμοι, αυτό είναι για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι αλλά και πιο θεραλέοι στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε αυτές τις υποδομες Συγγνώμη. Δυο-τρία θέματα που δεν ακούσαμε και θεωρώ σημαντικά είναι τα εξή. Ε, Είχαμε συζητήσει για την αλλίωση των στοιχείων των ε, ε, μετρητών, των ε, χιλιομετρητών. Για μας και για μένα αυτό έχει πολύ μεγάλη σχέση και με την ασφάλεια. Κανείς δεν αυξάνει αυτές τις ενδείξεις εθελοντικά, πάντα μειώνονται και αλλοιώνονται. Υπάρχει το σύστημα ΚΑΠ, υπάρχουν ε, και τεχνικές λύσεις άλλες που θα πρέπει να το καθιστούν αυτό αδύνατο. Για τις στατιστικές ε, σχέση με τα τροχέα, το είπε και ο συνάδελφος Κοχ, ότι συλλέγονται κάποια στοιχεία που βοηθούν και την έρευνα και την κοινοτομία αλλά και την ε, πρόληψη των δυστυχημάτων. Θα πρέπει να συλλέγουμε και άλλα στοιχεία όμως. Παράδειγμα, πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται λόγος για τα θύματα του κάψωνα. Το 2015 37 Παιδιά πέθαναν στι Πολιτείε επειδή τα ξέχασαν στο αυτοκίνητο μέσα σε κάψωνα. Στην Ευρώπη δεν μαζεύουμε τέτοια στοιχεία. Η προστασία των δεδομένων δεν αφορά μόνο την ιδιωτική ζωή, αλλά και γενικότερα την ασφάλεια. Για να έχουμε αποδοχή στα μάτια του κόσμου θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων. Από hackers, από εχθρική ε, χειραγώγηση ε, των στοιχείων και από πρόσβαση στα στοιχεία εξ αποστάσεως. Ε, πολύ σημαντικά και πολύ χρήσιμα αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι και νομίζω ότι είναι καλή αυτή η έκθεση πρωτοβουλία τη Επιτροπής μα. Και πάλι λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μεγαλύτερε φιλοδοξίε. Ευχαριστώ πολύ. Merci à vous. Ευχαριστώ, κύριε Άντερσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη έκθεση. Ακριβώς και λόγω όλων των πρωτοβολιών που έρχονται για θέματα ασφάλειας των φορτηγών και για θέματα του πακέτου οδικών και σιδεροδρομικών μεταφορών. Και χαίρομαι και για τα σχόλια που έχετε ε, εκφράσει. Στηρίζω την ανάγκη να μειωθούν οι τυφλές γωνίες ε, για τους οδηγούς των ε, φορτηγών και βαρέων οχημάτων και πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι. Όμως η παράγραφος 20 για τα θέματα άμεσης όρασης θα πρέπει να ενισχυθεί. Κύριε Κόχ, καταλαβαίνω ότι είσαστε επιφυλεκτικός και δεν θέλετε να βάλετε συγκεκριμένες καταληκτικές προθεσμίες, όμως μόνο μια εξαίρεση να προβλέψουμε γι' αυτό παρακαλώ και συμφωνώ και με αυτό που είπε ο κύριος Ζλατόφσκι. Είναι κρίσιμη και απόλυτη σημασία να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τα πολύ βαρέα οχήματα, τα βαριά, τα μεγάλα φορτηγά, όχι μόνο εντό άστεως αλλά και σε γενικές γραμμές γενικότερα. Για τα ελαστικά η ασφάλεια των ελαστικών είναι ένα θέμα που έχει παραμεληθεί συχνά σε αυτή τη συζήτηση. Θα υποβάλω ορισμένε τροπολογίε ω προ αυτό και ω προ τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πίεση των ελαστικών. Υπάρχουν διεθνή πρότυπα και νομίζω ότι θέλετε και θα ήταν καλό να τα αναφέρετε. Η Επιτροπή μας γνωρίζει πολύ καλά πόσο πολύ έχουμε συνεργαστεί και έχουμε δουλέψει για τις διαστάσεις, τα βάρη και τα μεγέθη. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί κατά πόδας και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δράση μας έτσι ώστε τα θέματα των διαστάσεων και βαρών να εξεταστούν με πιο γρήγορο ρυθμό. Τώρα για το γενικότερο κανονισμό για τη γενικότερη ασφάλεια είναι κάτι που μας, τον έχουν, μας έχουν υποσχεθεί εδώ και πολύ καιρό. Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να υπογραμμίσει ότι δεν πρέπει να γίνουν περαιτέρω καθυστερήσεις για αυτή την αναθεώρηση. Συμφωνώ με τον κύριο Κράμε και για τα αυτόματα συστήματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικά να έχουμε ισχυρή προσέγγιση. Να μην κλείνονται, να μην μπορεί κανείς να τα πενεργοποιήσει, εκτός από πολύ κατεξαίρεση της συνθήκης. Είτε πρόκειται για συστήματα αυτόματης πέδησης ή άλλα είδους συστήματα δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτό ο εκάστοτε οδηγός να μπορεί να τα απενεργοποιεί κατά βούληση. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες και όλους όσοι συμμετείχαν στην πολύ καλή συζήτηση που οδήγησε σε αυτό το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ, Σέντερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κόχο για το ενδιαφέρον που παραδοσιακά καλλιεργεί και την ε, πολύ προχωρημένη σκέψη του, διότι μας δίνει νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για να ενισχύσουμε έτσι περαιτέρω την ασφάλεια των οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι προχωρούμε εν αναμονή και μας ε, ενοχλεί το γεγονός ότι πράγματι καταφέραμε να βελτιώσουμε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οχήματα και να λύσουμε τα προβλήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας, δηλαδή να, σε κάποιο βαθμό να βελτιώσουμε τα τεστ σε ό,τι έχουν να κάνουν με την πρόσκρουση με ε, πεζούς και ποδηλάτες. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε και θα πρέπει να το πράξουμε, όμως υπάρχει μια μικρή ασυνέπεια. Τι εννοώ, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε εξετάζουμε να ενισχύσουμε περισσότερο την ασφάλεια των οχημάτων και κυρίως τον, την ασφάλεια των επιβατών τους, ενώ αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι ότι έρχονται συνεχώς όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένα οχήματα. Άρα, από τη βιομηχανία. Άρα η αλληλεπίδραση, η διεπαφή ε, μεταξύ οχημάτων και των χρηστών αυτού αλλά και των χρηστών του δρόμου όπου κινείται το όλο και πιο αυτοματοποιημένο όχημα, ε, οι χρήστες είναι πεζοί, ποδηλάτες και άλλοι, ε, αυτό δεν το έχουμε ακόμα συζητήσει αρκετά. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες σε αυτό εστιάζουν την προσοχή τους για να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Είναι όλο και πιο επιθετικές στο σχεδιασμό, όλο και πιο ψηλά τα οχήματα, όλο και πιο τετραγωνισμένα όλο και πιο ατσάλιτα αν θέλετε, λες και πρόκειται να μπουν σε ένα ε, νέο είδους αστικό πόλεμο. Ε, και απ' την άλλη προσπαθούν να σεβαστούν όλο και περισσότερο τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Ε, βασικά κείμενα, όπως η έκθεση Μαρκόφ για την ασφάλεια των υποδομών, που παρέμεινε σε θελούσια βάση στα κράτη-μέλη. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θελήσαμε να έχουμε εξωτερικούς ελεγκτές υποχρεωτικούς και κανόνες εξωτερικούς υποχρεωτικούς. Και θα πρέπει, αν τα οχήματα τελικά καταλήξουν να είναι πλήρως ε, αυτοματοποιημένα, τότε σίγουρα οι κανόνες και ο έλεγχος πρέπει να είναι όσο να το περισσότερο εξωτερικός, ανεξάρτητος και υποχρεωτικός. Και τελικά σταματήσαμε στα μισά του δρόμου. Δεν καταφέραμε αυτά να τα κάνουμε υποχρεωτικά. Αλλά και τις κυρώσεις δεν τις καταφέραμε να τις κάνουμε υποχρεωτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και το Συμβούλιο ακολούθησαν το Κοινοβούλιο, παραδέχθηκαν ότι ανάγκη να έχουμε πρότυπα και κανόνες που από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά από τη στιγμή που έχουν να κάνουν με παραβάσεις που αναγνωρίζονται παντού ως παραβάσεις και ε, με πράξεις που ε, πλήττουν την οδική ασφάλεια. Είναι αυτά στοιχεία λοιπόν με αυτά τα δεδομένα ε, είναι ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και πρέπει να λυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια θα πρέπει να περιλαμβάνει μία παράγραφο που να έχει να κάνει με την ασφάλεια των υποδομών και τη συμπεριφορά, άρα παράβαση, αναγνώριση παράβασης και κύρωση, τιμωρία των εκάστοτε χρηστών. Και θα πρέπει να υπάρχει και ένα διοικητικό σκέλος που έχει να κάνει με όλα αυτά στα οποία έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο για τους τραυματίες, όχι μόνο τους τραυματίες καθ' αυτούς, αλλά και για τις επίγουσες, τις πρώτες βοήθειες. Πώς θα προετοιμαστούμε, πώς θα προετοιμάσουμε με, ε, τις πρώτες βοήθειες με τη βέλτιστη δυνατή τεχνολογία, μέσα σε ένα αποδεκτό πλαίσιο δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε εξαιρετικά γρήγορη ανταπόκριση από πλευρά των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών σε περίπτωση οδικών ατυχημάτων. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Merci beaucoup. Monsieur Wim van den Kamp, Ευχαριστώ κύριε Βίμ Βαντενκάμπ. Ευχαριστώ πρόεδρε πολύ. Και τον Τίτερ Κόχ για το σχέδιο έκθεσή του. Καταρχά θα ήθελα να συμφωνήσω και με τη δική σας συναισθηματική έκκληση εγώ είμαι τρία χρόνια τώρα μέλος στην Επιτροπή Μεταφορών και κάθε μήνα συζητούμε για τους 22.000 νεκρούς ετησίως που έχουμε. Και αν δεν προσέξουμε θα το συνηθίσουμε κιόλας. Ζήσαμε τη Μοσούλη, ζήσαμε τη Συρία και στην Ευρώπη Έχουμε κάθε χρόνο 22.500 νεκρούς στην άσφαλτο. Αυτά ο κόσμος πώς τα καταλαβαίνει. Έχουμε την καταπληκτική διακήρυξη της Μάλτας που δεν αλλάζει τίποτα. Κάθε μέρα δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Μήπως θα πρέπει να μας απασχολήσει μια διαφορετική στρατηγική επικοινωνίας και ρωτώ και τον Τίτερ Κόχ. Δεύτερη ερώτηση, Πρόεδρε. Εγώ κατάλαβα ότι η έκθεση αυτή έχει να κάνει με την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Ε, ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων. Καμία σχέση με πεζούς, καμία σχέση με ε, την ασφάλεια την οδική γενικότερα. Έτσι, εν μέρη μόνο με τις υποδομές και χρειάζεται προσοχή να μην το κάνουμε εδώ χριστουγεννιάτικο δέντρο. Να βάλουμε όλο το ευκολόγιο για την οδική ασφάλεια στην έκθεση του Ντίτερ. Γιατί είναι εκτός τόπου αυτά. Εγώ θα επικεντρωθώ μόνο στα τεχνικά στοιχεία. Και όντω έχει σχέση ε, και με αυτό που είπε η Λούση Άντερσον για την τυφλή γωνία στους καθρέφτες. Επίσης τα φορτηγά, ε, η πίεση των ελαστικών ε, αυτό ελέγχεται αυτόματα πάνω κάτω. Και επίσης να μην κάνουμε να μην υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίηση αυτών των συστημάτων. Με την κυρία Σένα Λόβα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ κάναμε την έκθεση για το e-call και ένα συνάδελφος από την Άλτε ήθελε να απενεργοποιείται. Γιατί ε, ε, ξέρω εγώ, μπορεί να είχε καμιά φιλενάδα και να μην ήθελε να τον εντοπίζουν που βρίσκεται, αλλά ήθελε, μπορεί να το απενεργοποιεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να το κάνουμε τότε. Δεν είναι καλή υπηρεσία αυτή στους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμπ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σίμονς για λίγα λεπτά από την ΟΚΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εμείς 20 χρόνια το συζητάμε στην Επιτροπή την ΕΟΚΕ, το θέμα της οδικής ασφάλειας και η ε, βάση μας ήταν η γνωμοδότηση για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο 2011-2020. Και στο πλαίσιο αυτό ε, είδαμε και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ελέγξαμε. Ε, και με βάση αυτή κάναμε την γνωμοδότησή μας. Πού οδήγησε αυτό. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν. Απλώς να τονίσω μόνο μερικά πράγματα. Η έκθεση του κυρίου Κοχ περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρότασή Γι' αυτό εγώ για να μην μακρηγορώ δεν θα επεκταθώ. Θα υπογραμμίσω μερικά μόνο σημεία που θεωρούμε έτσι πιο σημαντικά και εξέχοντα. Στην έκθεση του κυρίου Κοχ λέει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ζήτημα των υποδομών εκεί θα πρέπει λίγο να σταθούμε. Κάναμε μια πρόταση, την οποία κάναμε και στο παρελθόν. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, κάνουν χάρτες με τα μελανά σημεία και να δημοσιεύονται που είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία για δυστυχήματα. Αυτή η πρότασή μας δεν ε, ευδοκίμησε πάρα πολύ. Στο Βέλγιο όμως τι συμβαίνει ε, μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιος χάρτης και διαδραστικός. Να έρχεται το κοινό ε, και να έρχονται και οι περίοικοι και να αντιδρούν και να λένε που γίνονται τα διάφορα δυστυχήματα. Και όταν θέλει το κράτος ή η πολιτική να αντιδράσουν, θα βλέπουν και τις αντιδράσεις των πολιτών. Γιατί όταν έρχονται οι πολίτες ε, και στο επισημαίνουν και πότε θα φτιάξει αυτή τη διασταύρωση να σταματήσει να σκοτώνεται ο κόσμος, τότε μπορεί να το καταλάβουν και οι πολιτικοί. Ε, τι φταίει και ε, πού έχουμε ε, θανατηφόρα τροχέα ή πολύ βαρύς τραυματισμούς. Ελπίζω η πολυ βαρυς τραυματισμος Επιτροπή αυτό να το σημειώσει ως ιδέα και να το προωθήσει αυτό το θέμα των διαδραστικών καρτών των μελανών σημείων στην ε, ε, κυκλοφορία. Κάτι άλλο τώρα. Κάτι ακούω για τα φορτηγά, ότι είναι υπεύθυνα για τα περισσότερα δυστυχήματα. Δεν θα το αμφισβητήσω και πιστεύω ότι δεν ισχύει πάρα πολύ αυτό. Σε διάφορα κράτη υπάρχουν συστήματα και προγράμματα που εφαρμόζονται όχι στις πόλεις, αλλά σε δρόμους, εθνικές οδούς και αυτοκινητοδρόμους. Και ε, έχει μειωθεί και ο αριθμός των φορτηγών που κυκλοφορούν. Από, από τρία, ας πούμε, έχουν γίνει δύο. Το τελευταίο είναι η προστασία των ε, ποδηλατών και των πεζών. Ουσιαστικά η λύση εδώ είναι πραγματικά υποδομές και επίσης τα οχήματα να έχουν συστήματα ανείχνευσης για να μπορούν να ανοιχνεύουν τους ε, πεζούς και τους ποδηλάτες. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και διάφορα συστήματα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω επίσης να κοιτάξετε και ε, τα δίκυκλα και τις μοτοσικλέτες. Ο κύριος Βαντενκάμπ είναι πιο έμπειρος από μένα. Αλλά αυτή είναι μια ε, ανυπεράσπιστη κατηγορία, οι μοτοσικλετιστές. Εγώ κάνω πολύ συχνά τη διαδρομή Αμβέρσα Βρυξέλλες που έχει πάρα πολλά αποτυλιαρίσματα και ε, ε, τα μηχανάκια σε ξεπερνάνε και έρχονται ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Αυτό επιτρέπεται ε, στο Βέλγιο, σε άλλες χώρες απαγορεύεται, αλλά απέρνουν μαζί τους και συμπαρασύρουν πόρτες, παράθυρα, καθρέφτες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, θα παρακαλούσα να σκεφτούμε και αυτή την κατηγορία χρηστών που χρειάζονται προστασία, που είναι ε, τα δίκυκλα με μηχανή. Σα ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, εγώ θα ήθελα να θυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορούμε και δεν, και δεν θα μείνουμε ε, αδρανείς μπροστά σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Όλοι οι φορείς, και το λέω αυτό που με ιδιαίτερη βαρύτητα, όλοι οι φορείς οφείλουν να ευαισθητοποιηθούν, να στηριχθούν, να πλαισιωθούν, αλλά και να τιμωρηθούν όταν χρειάζεται. Όταν λέω ότι είναι σοβαρό θέμα, είναι σοβαρό γιατί πρόκειται για ζωές. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμίζουμε ότι η ασφάλεια στους δρόμους θα πρέπει να καταστεί δικαίωμα για κάθε πολίτη όπου και αν βρίσκεται στην Ευρώπη. Non, suite à Τώρα, σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα λοιπόν, και ευχαριστούμε κύριε Κόχα για την έκθεσή σας, το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα τονίσετε το θέμα της ε, χρηματοδότησης των ποιοτικών οδικών υποδομών Δηλαδή πώς ε, θα μπορέσουμε να ασφαλίσουμε τους δρόμους μας ε, καλύτερα ε, από αύριο, πώς θα βελτιωθούν οι τεχνικοί ελέγχοι κταίω, πώς και αν υπάρχουν και πώς θα χρησιμοποιηθούν τα γεφείς υπηρεσίες όπως το e-call, αλλά είναι και το θέμα της επιμόρφωσης. Θα εγγυηθείτε και θα πρέπει αυτό να το δούμε και ω συνέπεια από έχω αυτής έκθεσης. Θα εγγυηθείτε μια ε, ισχυρή και διαρκή δράση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η οποία είναι απαραίτητη ε, αύριο είτε πρόκειται για αποδηλάτες είτε για πεζούς θα πρέπει να τους εγγυηθούμε δικαιώματα για να μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας δώσω το λόγο στον κύριο Ράουερτ Έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη στις πλάτες σας, στους ώμους σας. Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην ακούμε πια λόγια και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες συνέργειες. Thank you, Madam Chair. And, uh, on σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της DigiGrow ε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, διότι ε, αντικατοπτρίζει τα σημεία κλειδιά που και η Κομισιόν έχει εντοπίσει. Επίση τονίζει αρκούντος το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων. Έχουμε φυσικά δράσει σε επίπεδο τη Ένωση που είναι για μα. Ε, Επίση αυτό μοιράζεται ανάμεσα σε, και σε άλλου συναδέλφου άλλων ε, γενικών διευθύνσεων, αλλά πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και από του κατασκευαστέ οχημάτων. Και όπω είπα, Επίσης αναγνωρίζουμε και ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια θέματα από διάφορα τμήματα της Επιτροπής. Αλλά εγώ είμαι σήμερα εδώ για τα θέματα ασφάλειας των αυτοκινήτων και βεβαίως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα και σε εθνικό επίπεδο και αν μιλάμε για παράδειγμα για την επιβολή ή για τη βελτίωση των υποδομών, αυτά όλα αναγνωρίζονται και όσον αφορά κάποια ζητήματα πρόσβασης στα στοιχεία, οι συνάδελφοι από την DG Move και την DG Just θα αποφασίσουν για να πώς θα προχωρήσουν σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να πούμε ειλικρινά ότι διστάζουμε να το καταστήσουμε αυτό μέρος της διαδικασίας έγκρισης τύπου, γιατί Μιλάμε για ασφάλεια οχημάτων και για μέτρα ασφάλειας επί των οχημάτων και αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Αρκετοί ομιλητές, οι περισσότεροι, ε, συμφωνούν με τον εισηγητή και είμαι ευτυχής που βλέπω ότι υπάρχει τέτοια ομόνια και εμεί θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι. Στο πλαίσιο του Horizon ιδιαίτερα καινοτόμα μέτρα έχουν προβλεφθεί. Διστάζω να τα πω ε, μέτρα, αλλά πάντως ε, συσκευές και ε, οι οποίες ήδη έχουν αποδειχτεί ασφαλείας και που θέλουμε να γίνουν πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων. Επίσης, σκεφτόμαστε διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διάφορες ε, κλάσεις αυτοκινήτων, ώστε να έχουμε μια καλή στρατηγική όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις τυφλές ε, γωνίες στα φορτηγά. Για φορτηγά ε, κυκλοφορούν μόνο στους αυτοκινητοδρόμους ενώ άλλα κυκλοφορούν και μέσα στις πόλεις όπου κάνουν παραδόσεις και είναι πολύ πιο επικίνδυνα για τους πεζούς και τους ε, ποδηλάτες. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα του βάρους και των διαστάσεων και της σχετικής οδηγίας. Αυτό θέλουμε με συνεπή τρόπο να το αντιμετωπίσουμε, ώστε να έχουμε μέτρα που δεν θα είναι αντίθετα μεταξύ τους, αλλά που θα είναι ε, συμπληρωματικά. Και για την ε, περιορισμό της ταχύτητας. Ειδικά για αυτό το σημείο μπορούμε να σας πούμε ότι σκεφτόμαστε και μια συνεργασία με τον οδηγό, δηλαδή όχι μόνο ε, σφυρίγματα, αλλά πραγματικά να ε, μπορεί να υπάρξει παρέμβαση στον γκάζι του αυτοκινήτου για να περιοριστεί η ταχύτητά του αυτόματα. Και βεβαίω κάτι ακόμα που θέλω να τονίσω, ότι οι ευάλωτοι χρήστες των δρόμων περιλαμβάνονται ε, στις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε. Επίσης θα αναθεωρήσουμε την ε, ε, οδηγία περί ασφάλειας των πεζών, το κανονισμό μάλλον περί ασφάλειας των πεζών, ε, ε, εκτός από τη Γενική Οδηγία Ασφάλειας. Και επίση την ειδοποιήσει των αυτοκινήτων για πεζούς ώστε να υπάρχουν λιγότεροι τραυματισμοί. Και προσβλέπουμε συνεργασία, στενή συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Vous parlez d'un paquet global. Vous avez un... Κάτι για ένα ε, συνολικό πακέτο. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, δεν κατάλαβα. Thank you. That's a fair question. Ευχαριστώ. Μάλιστα, για την ώρα προετοιμάζουμε την ε, μελέτη αντικτύπου, γιατί βεβαίω αυτό που τονίζει η έκθεση είναι ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά ως προς το κόστος και όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και τώρα δουλεύουμε πάνω σε αυτήν θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να είμαστε Ελπίζουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε την πρόταση της Κομισιόν μέχρι την άνοιξη του επόμενου χρόνου. Και εκεί θα περιλαμβάνονται ειδικά τα μέτρα τα οποία θέλουμε να εισάγουμε. Donc, vous êtes tous témoins, Όλοι είστε μάρτυρες αγαπητοί μου συνάδελφοι. Άνοιξη της επόμενης χρονιάς θα είναι προτεραιότητα για την Κομισιό. Θα πρέπει βεβαίως αυτό, αυτή η προτεραιότητα να υιοθετηθεί πριν το τέλος της θητείας. Και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κόχ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε περάσει κατά μισή ώρα το πρόγραμμά μας. Δεν θέλω να απαντήσω σε όλους τους ομιλητές, ούτε σε όλα τα επιχειρήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που τονίζετε και τη σημασία της έκθεσης αυτής για τους πολίτες, ε, τους Ευρωπαίους που πραγματικά περιμένουν να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι απτό, χειροπιαστό, καλό για τους ίδιους. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχετε δει και αυτή που λέτε ότι δεν θα πρέπει να προστατεύουμε περισσότερο τους επιβάτες του αυτοκινήτου του οχήματο, να μην έχουμε τροχιά με νεκρούς ε, στο αυτοκίνητο του τάδε κατασκευαστή, αλλά μας ενδιαφέρουν όλοι οι χρήστες του δρόμου, νέοι, ε, ηλικιωμένοι, πεζοί, ποδηλάτες, άνθρωποι με αναπηρίες. Όλο τον κόσμο θέλουμε να προστατεύουμε και να ε, μας απασχολεί. Βεβαίως, πάντα τίθεται το θέμα του κόστους. Ε, που πρέπει να αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν πολλά συστήματα αλληλοσυμπληρούμενα που έχουν τους ίδιους ας πούμε αισθητήρε. Όταν έχεις ένα σύστημα στο αυτοκίνητο το να επεκταθεί σε ένα δεύτερο ή τρίτο δεν είναι τόσο ακριβό και επίσης η μαζική παραγωγή και ε, εγκατάσταση στα αυτοκίνητα μειώνει και το κόστος ε, ριζικά και μαζικά. Άρα αυξάνεται και η αποδοχή ε, του πληθυσμού, που είναι και η άλλη όψη του νομίσματος. Η μία όψη είναι η υποχρεωτική νομοθεσία, που ορισμένοι το ζητούν και σου λένε θέλω και να το πληρώσω. Η έκθεση μου είναι έκθεση πρωτοβουλία. Αυτό που με ενδιαφέρει να πούμε τι θέλουμε. Τώρα όλες οι λεπτομέρειες, προθεσμίες κλπ. Ε, θα τις δούμε αργότερα ε, στον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια. Δηλαδή, και ποια ποια συστήματα παρακολούθησης, πότε θα χρησιμοποιούνται ή ένα καλύτερο σύστημα για ε, την πέδηση. Δηλαδή να μην είναι μείωση ένας κόφτης ταχύτητας κατά 20 χιλιόμετρα, αλλά να κοκαλώνει το αυτοκίνητο επιτόπου. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε. Είναι λεπτομέρειες το θέμα της απενεργοποίησης των συστημάτων αυτών και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και πρέπει να το συζητήσουμε διότι αυτό το, λένε διάφοροι, όχι κατασκευαστές, αλλά ΜΚΟ, λέσχες αυτοκινήτου και λοιποί, θέλουν να μπορούν να τα κλείνουν αυτά τα συστήματα. Εγώ είμαι αντίθετος να το συζητήσουμε, να δούμε τι θέλουμε ως πολιτικοί να νομοθετήσουμε. Τελευταίο θέμα, το ενόπνευμα. Ε, εγώ είμαι από την Ανατολική Γερμανία που απαγορευόταν απολύτως να πιείς και να οδηγήσεις. Μηδέν της χιλής ήταν. Και ε, αυτό δεν περνάει παντού στην Ευρώπη και ορισμένοι επιστήμονες λένε ακόμα και αν πιείς ένα μιλίτι, ας πούμε κάτι που να έχει ένα ε, πολύ μικρό αλκοόλουχο βαθμό, μπορεί να δώσει θετικό αποτέλεσμα στο αλκρότες. Για τους αρχάριος πάντως για μένα και τους επαγγελματίες οδηγούς θα πρέπει να απαγορεύεται απολύτως, τα υπόλοιπα τα συζητάω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόχ. Καταληκτική προθεσμία υποβολής τροπολογιών 14 Ιουλίου στις 11 η ώρα. Προχωρούμε με το ψήφισμα για την Πολυμερή Συμφωνία για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Η συγητής είναι ο κύριος Ρόμπερτς Ζήλε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια πολυμερή συμφωνία που καλύπτει τα χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, την Νορβηγία και τα ε, έξι κράτη της Βαλκανικής, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η Φιρόμη, η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Αλβανία και άλλες χώρες. Ε, όλα αυτά ξεκίνησαν το 2016 και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ολοκλήρωση της συμφωνίας και υπερψήφισε την έκθεση της κυρίας Λίχτενμπέργκερ τον Απρίλιο του 2007, λέει μιλητής. Η διαδικασία κύρωσης ολοκληρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη από το 2006-2007 μέχρι το 2014 και τον Νοέμβριο του 2015 παρουσιάστηκε τροποποιημένη πρόταση για την απόφαση του Συμβουλίου να συνάψει αυτή τη συμφωνία λαμβάνοντα υπόψη τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Βουλγαρία και το γεγονό ότι Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία είχαν γίνει εντωμεταξύ πλήρη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τώρα αυτή τη νέα διαδικασία και με αυτή τη συμφωνία οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, δεσμεύονται ότι θα διγραμμίσουν την ομοθεσία τους με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε όλα τα θέματα των μεταφορών και κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με ασφάλεια και επάρκεια ε, στις μεταφορές, στις εναέρειες μεταφορές. Ε, πριν από 10 χρόνια ξεκίνησαν όλα αυτά, το 2006 παραπάνω από 10 χρόνια και είχαμε προσωρινείς ρυθμίσεις για τις χώρες που είναι εταίρημα στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Και έτσι αυτή η διαδικασία άνα ε, βήμα ε, έχει προχωρήσει για να υπάρχει ευθυγράμμιση με τους κοινωτικούς κανόνες και πρότυπα. Άρα όλες αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρώνονται και τα προαπαιτούμενα από τις χώρες εταίρους μας, ειδικά για τους κοινούς κανόνες ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τη διαδικασία σύγκλησης και τον τρόπο ε, εφαρμογής των μέτρων για την ασφάλεια και δίδει τεχνική βοήθεια στις χώρες εταίρους. Αναλόγως και με τις ανάγκες των χωρών αυτών επιτόπου και ο αρμόδιος επίτροπος θα παρουσιάσει έκθεση προόδου για κάθε χώρα εταίρο μας. Είναι θετικές οι συστάσεις για την σύναψη της συμφωνίας, για την ολοκλήρωση αυτής. Εμείς μπορούμε να την απορρίψουμε, να την ε, εγκρίνουμε και γι' αυτό στην έκθεσή μου καταλήγω στο συμπέρασμα ότι πρέπει να την εγκρίνουμε τη συμφωνία. Η καταληκτική, τροποθεσία, ε, καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι πολύ μικρή. Σήμερα μέχρι τις 7 το βράδυ μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες και αύριο το πρωί θα γίνει ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ζήλε, σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντέλη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα για την υποβολή τροπολογιών, αλλά εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που έχουμε φτάσει σε αυτό το καταληκτικό στάδιο μετά από δέκα και πλέον έτη. Όλα ξεκίνησαν το 2006, όπως πολύ σωστά είπε ο εισηγητής. Η κύρωση της συμφωνίας έγινε πριν από τρία χρόνια. Εν τω μεταξύ είχαμε νέα προσχώρηση, είχαμε και νέα συνθήκη Επομένως, ε, έχει έρθει η στιγμή να τροποποιήσουμε την ε, διακρατική πολυμερία αυτή συμφωνία και τη στηρίζει αυτή τη συμφωνία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνοντας την ε, έκθεση του κυρίου Ζήλε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ των φιλελευθερών ο κύριος Ράντος. Υποστηρίζουμε τη συμφωνία αυτή. Δεν υπάρχει τίποτα επίμαχο ή αμφισβητούμενο. Απλώς ε, ε, υπεγράφει το 2006 η συμφωνία αυτή. Εδώ πρόκειται για την ενσωμάτωση των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στη συμφωνία αυτή ε, και την ένταξή τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτή η διαδικασία βαίνει με ταχύτερους ρυθμούς από ότι η πολιτική ολοκλήρωση. Ε, στον τομέα των μεταφορών και στις αερομεταφορές ε, έχουμε αρχίσει αυτή την προσπάθεια ήδη από το 2006 και μετά την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, ε συνορεύουν, περικυκλώνονται ουσιαστικά από ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να ενταχθούν και να ενσωματωθούν σε όλους τους κλάδους των μεταφορών, όχι μόνο για τις εναέρειες μεταφορές δηλαδή, αλλά και ε, αλλού. Και σε άλλα θέματα περιβάλλον, οικονομία γενικότερα. Ευχαριστώ κύριο Στέιλορ. Α, δεν θέλετε. Okay. No. Madame... Ε, ε, κυρία Ορνοτού, παρακαλώ. Merci, merci, Madame Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι πώς η Επιτροπή μας μπορεί να δώσει μια σύσταση στο Συμβούλιο από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα αξιόπιστο στοιχείο και καμία αξιόπιστη πληροφορία. Η μόνη σοβαρή μελέτη είναι η μελέτη που έχει αναθέσει η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και είναι του 2013. Οι συμφωνίες που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας δεν έχουν ως αποτέλεσμα ε, αύξηση της κυκλοφορίας, ούτε επηρεάζουν ιδιαίτερα την ε, κυκλοφορία και την κίνηση. Ωστόσο, άλλες χώρες έχουν ανάπτυξη του εναέρι, της ενιάρης κυκλοφορίας παράλληλη και ε, παρεμφερή με τα ευρωπαϊκό, με τα ευρωπαϊκά νούμερα. Όλα αυτά αποτελούν τροχοπέδι για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του, εθνικού, του ευρωπαϊκού και εκτιμένου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την επιχειρηματολογία της σε μια μελέτη που έγινε από μπούς και λοιπούς. Και σύμφωνα ε, με αυτή τη μελέτη ο απολογισμό για τα Δυτικά Βαλκάνια θα είναι καλό, όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτό και αν σφάλω δεν έχει δημοσιεύσει αυτή τη μελέτη, αυτή την έκθεση. Θα ήθελα κύριε Σιγητά και θα σα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μα διευκρινίσετε όλα αυτά τα θέματα και κυρίω σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια ε, και την ε, επάρκεια απρόσκοπτη ευρωπαϊκή κυκλοφορία, εναέρια κυκλοφορία. Θα Πρέπει να πούμε ότι τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπεται να διαλέξουν τους τρόπους και τις συνθήκες διαχείρισης των υπηρεσιών εναέριων μεταφορών και αυτό ε, είναι μέρημνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι παρεμποδίζεται η εθνική κυριαρχία, υπονομεύονται οι εθνικές υπηρεσίες, τελικά ε, χειροτερεύουν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι εξαιρετικά δυστυχές όλο αυτό. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το control δεν είναι αρκετή εγγύηση. Είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της μελλοντική προσχώρησης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική προσχώρηση και ε, όπως γνωρίζετε η πολιτική μου ομάδα δεν συμφωνεί με αυτό ε, δεδομένη της καταστροφικής προσχώρησης των προηγουμένων χωρών που έγιναν μέλη. Θα ήθελα ορισμένε διευκρινήσεις κύριε Σιγητά, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Άλμπερτον είναι εδώ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Μετά από αυτά τα ερωτήματα μπορείτε να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει ε, τη στήριξη του εισηγητή η οποία θα μας επιτρέψει, όπως εξήγησε και ο εισηγητής, να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε πλήρως μια συμφωνία που υπογράφει και πριν από 10 χρόνια, μια συμφωνία που θα μας επιτρέψει να ε, δώσουμε στις χώρες όλα τα ωφέλη. Ε, οι χώρες που θα υποφεληθούν από αυτή τη συμφωνία θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τον ενάριο τους χώρο. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις θέλω να σας πω ότι αυτό σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή η νομοθεσία για την ασφάλεια, για την επάρκεια της εξυπηρέτησης, θα ενσωματωθούν πλήρως και θα εφαρμόζονται πλήρως σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν και προσχωρούν στη συμφωνία. Άρα η συμφωνία θα επιτρέψει την ύπαρξη ίδιων προτύπων. Τα ίδια στάνταρ, τα ίδια πρότυπα θα εφαρμοστούν σε όλες τις εμπλεκόμενες και συμμετέχουσες χώρες εξού και ο κοινός ευρωπαϊκός εναέριος χώρος ε, βγάζει νόημα και είναι λογικό εκεί η ύπαρξή του. Οι χώρες αυτε, καθ' αυτές έχουν σημειώσει αρκετή πρόοδο ε, χρόνο με το χρόνο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εμπειρογνώμονες της ε, ε, Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας αξιολογούν κάθε χρόνο την πρόοδο που σημειώνουν οι συμμετέχουσες χώρες και η πλήρης ολοκλήρωση της συμφωνίας θα επιτρέψει να μεταφραστεί αυτή η πρόοδος ε, με νομικούς όρους, να κατοχυρωθεί αν θέλετε νομικά και θα έχουν οι χώρες αυτές πρόσβαση στην εσωτερική αγορά. Η μεταβατική περίοδος μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί η συμφωνία δεν είχε τεθεί σε ισχύ. Θα προσδιοριστούν αυτά άπαξ και ολοκληρωθεί και συναυθεί η συμφωνία και όπως προβλέπεται στην συμφωνία καθ' αυτή όλα τα προαπαιτούμενα ορίζονται ανά χώρα. Γι' αυτό και δηλώνεται ότι το γεγονός ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ε, είναι, μέλη του Eurocontrol και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η ΚΑΟ, αυτό ε, ε, δεν σημαίνει αλληλοεπικάλυψη. Το και ευρωπαϊκό κεκτημένο που υπάρχει στη συμφωνία θα πρέπει να εθετηθεί πλήρω από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρο και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριο Ζήλε παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Να σχολιάσω ε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να στηρίξουμε ή να, στηρίξ, να μην στηρίξουμε νέες τροπολογίες. Αν έχετε τροπολογίες μπορείτε να τις υποβάλλετε μέχρι τις 7 το βράδυ. Εάν δεν τη στηρίξουμε θα είναι βλάβη σε μία αγορά 500 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 36 χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία από την Ενωμένη Ευρώπη, διότι αυτές οι χώρες ήταν υποψήφιες όταν συνήφθηκε η συμφωνία, αλλά τώρα είναι πλήρη μέλη. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζήλια. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των ε, τροπολογιών. Απόψε μέχρι τις 7 έχετε περίπου ένα δίωρο. Συνεχίζουμε λοιπόν και προχωρούμε στην διεθνή διαχείριση των Οκεανών, ένα πρόγραμμα για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων της αηφόρου ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Είναι μια γνωμοδότηση πάρα πολύ καλή για τους στόχους της διάσκεψης των μερών 21 για το κλίμα. Η συγκήτρια δεν είναι εδώ και ο κύριος Βιμ Βαντενκάμπ θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι ζητάει συγγνώμη η συγγήτρια η κυρία Κλάουδια Μοντέρο. Κανονικά στην ημερήσια διάταξη, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης, ε, το θέμα της προβλεπόταν αύριο και άλλαξε τώρα και ήρθε σήμερα. Διαβάσατε ότι προσπάθησε ε, να συμπεριλάβει διάφορα στοιχεία των ωκεανών. Ο ωκεανός είναι χρυσός, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος, όπως είπατε κι εσείς. Και χρειάζεται βελτίωση η θαλάσσια κυκλοφορία που είναι και μεγάλη στους ωκεανούς. Οι ωκεανοί έχουν μια μεγάλη οικονομική προοπτική και διάσταση και για τις μεταφορές, γιατί πολλά αγαθά μεταφέρονται δια θαλάσσης και αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι τα κράτη-μέλη πριν ε, τις 31 Μαρτίου του 2021 θα πρέπει να έχουν κάνει τη θαλάσσια χωροταξία τους και να την έχουν ε, καταθέσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαφυλάξουμε και να διασώσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και ένα μεγάλο στοιχείο για την ασφάλεια. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα στη Μεσόγειο με τους πρόσφυγες που έρχονται με σκάφη και πώς συνεργάζονται οι οργανισμοί για την ασφάλεια στη θάλασσα, Frontex και το EFSEA Είναι προτεραιότητα αυτό και για την Κλάουντια Μοντέρο και δεν θα πρέπει να λησμονούμε, Πρόεδρε, την καινοτομία εδώ και την ψηφιοποίηση. Στη θάλασσα μπορούμε να έχουμε ακόμα περισσότερες εφαρμογές και της καινοτομία και της ψηφιακής ε, τεχνολογίας. Για το περιβάλλον, ε, θέλω λίγο την προσοχή σας για την οδηγία ε, για τις λιμενικές εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την θαλάσσια ρήπανση ε, αν εφαρμόζεται σωστά και η Κλάουδια εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμπεριλαμβάνει τον τουρισμό και τον αφαίρει στην εκθεσή της συγκεκριμένα στην παράγραφο 8 της σύστασης, ε, της νομοδότησης καλύτερα. Επαναλαμβάνω, οι ωκεανοί είναι ευκαιρία, απειλούνται, ε, έχει μεγάλη σημασία η ασφάλεια αλλά και ο τουρισμός. Αυτά εισαγωγικά εξ ονόματος της Κλάουντια Μοντέιρο. Ε, Ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο θα πάρουν οι σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία που δεν σας βλέπω. Εδώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Και για μένα η διεθνής ε, ε, θαλάσσια πολιτική είναι σημαντική για να έχουμε και πιο αποτελεσματική αλλά και πιο αηφόρο ε, κοινή χρήση των θαλασσών και των ωκεανών. Γι' αυτό καλωσορίζω την κοινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάτης εκπροσώπου και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κάποια σημεία ε, που είναι ουσιαστικά ε, για τη δική μας επιτροπή. Αυτό είναι η χωροταξία στη θάλασσα, οι θαλάσσιες, ε, γαλάζιες τεχνολογίες για την γαλάζια ανάπτυξη, ψηφιοποίηση ή ακόμα και ιδέα διεθνούς συνεργασίας για να, απο... Ε, να ξεφύγει η ναυσιπλοεία από την εξάρτησή της από τον άνθρακα. Εγώ είμαι σκιώδης συγγήτρια ε, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και θα ήθελα να ε, συμπληρώσω κάποια θέματα, θα κάνω και τροπολογίες. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε διεθνείς στρατηγικές αποτελεσματικές για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και άλλες ε, βλαβερές εκπομπές της ναυτιλίας. Θα πρέπει ο κλάδος να συνεισφέρει όσα το αναλογούν βάσει της Συμφωνίας των Παρισίων για την προστασία του ε, περιβάλλον θα πρέπει να απαγορευτεί στην ακτική τα σκάφη να ε, καίνε ε, βαρύ πετρέλαιο. θα πρέπει να δημιουργηθούν δυνατότητες έτσι ώστε να τηρούνται οι διεθνείς συμφωνίες και να επιβάλλονται και οι έλεγχοι. Αυτό αφορά ιδιαίτερα ε, αναψώμενες χώρες και μικρές νησιωτικές χώρες. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα απειλούνται από απόβλητα ε, από παράνομες ε, απορρίψεις ε, και καθαρισμούς δεξαμενών και από έλλειψη λιμενικών εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να έχουμε στρατηγικές και μέτρα που να είναι συγκεκριμένα και να ελέγχονται. Μόνο με τη βελτίωση της διαφάνειας, με σαφή επίρρηψη ευθυνών και υπεύθυνη στάση όλων θα έχουμε πρόοδο. Χαίρομαι για τη συνεργασία και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ, ο κύριος Δεμέσμακερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μοντέρο για το έργο της. Στις 8 Ιουνίου ήταν Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών και είδαμε ε, πόσο μεγάλη είναι η πίεση που απειλεί τους ωκεανούς. Βέβαια ε, και ε, είχαμε ε, εξαγριωθεί, εξοργιστεί. Αλλά μία μέρα οργής δεν αρκεί για να εφαρμοστεί το σημείο 14 της στρατηγικής για τους ωκεανούς. Ε, και για τον άνθρωπο είναι σημαντικές οι θάλασσες, σταθεροποιούν το κλίμα, απορροφούν ε, το 1 τέταρτο του διοξιδίου του άνθρακα και παράγουν οξυγόνο. Και φυσικά οι ωκεανοί παίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομία μας. Είναι πηγή ανανεώσιμης ενέργειας ε, συμμετέχουν και μεταξύ άλλων ε, διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο αλλά και τον τουρισμό. Και αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία ε, μας ενδιαφέρουν στη δική μας γνωμοδότηση και θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Το σύνολο της ανακοίνωσης και το σχέδιο έκθεσης ζυγήτριας μπορεί να είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Η ομάδα μου υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, για το διεθνές εμπόριο και τη διεθνή ε, μεταφορά επιφατών. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους για την ασφάλεια, για την αλεία, για το περιβάλλον, με σεβασμό στην επικουρικότητα. Με καλό συντονισμό ανάμεσα ε, στους οργανισμούς EFCA, EMSA και Frontex για να ε, χρησιμοποιούμε καλύτερα τις υφιστάμενες υποδομές και να αξιοποιούμε καλύτερα τις δυνατότητες. Επίσης υπάρχει και ο θαλάσσιος και παραθαλάσσιος τουρισμός ε, στην Ευρώπη ε, δημιουργεί 3,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και παράγει 183 δισεκατομμύρια ευρώ πλούτο. Θυμίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στην διαπραγματευτική εντολή για το πακέτο για τα απόβλητα ζητεί μείωση ε, στο μισό των απορρίψεων μέχρι το 30% μέχρι το 2025 και αξιόπιστη ε, μέθοδο μέτρησης. για να παρακολουθούμε και τι γίνεται με τα ε, πολύ μικρά σωματίδια που διαλύονται στους ωκεανούς και ρηπαίνουν και προκαλούν ε, βλάβες. Ε, τελικά οι ωκεανοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου στη γη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς δεν το συνηθίζω, αλλά θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο που αγωνίστηκε να πάρει αυτό το θέμα η Επιτροπή Μεταφορών. Γιατί είναι έκθεση Επιτροπής Μεταφορών, θα πρέπει να το γνωρίζουμε. Το 2007 ε, εφευρέθηκε η πολιτική για τη θάλασσα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη γαλάζια ανάπτυξη, για τη χωροταξία. Ήταν πάντα αρμόδια ε, η δική μας Επιτροπή. και κανονικά δεν ήταν θέμα τη Επιτροπή Περιβάλλοντος και επειδή αγωνίστηκε η πρόεδρό μας έχουμε συναρμοδιότητα. Ε, βέβαια γνωμοδότηση μα έδωσαν, αυτό δεν είναι αρκετό. Για τρία θέματα έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα και κάποιε άλλε αρμοδιότητε είναι κοινέ. Δυστυχώ δεν έχουμε την εισηγήτρια παρούσα και την ευχαριστώ. Είπε ε, ότι... Ε, νόμιζε ότι είναι αύριο το θέμα της. Κανονικά θα ήταν αύριο και άλλαξε. Ξέρω ότι η Κλάουντια είναι πάρα πολύ δραστήρια και κατάφερε σε 8 μέσα σημεία να κάνει, γιατί μια γνωμοδότηση πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομη, ε, έκανε τεράστια προσπάθεια για να τα συμπεριλάβει αυτά. Και είμαι βέβαια ότι και η δική μας γνωμοδότηση θα συμπληρωθεί και εγώ θα κάνω τροπολογίες, τα είπε και η κυρία Ρόντουστ και ο κύριος Δεμέσμακερ, και η συγγήτρια ίδια. Οι οικοκιανοί για το μέλλον της ανθρωπότητας ε, έχουν τεράστια κομβική σημασία και είμαι κράτοντα πεπισμένη γι' αυτό. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την ανάπτυξη των θαλασσών, των ε, ωκεανών και τι γίνεται και με ε, τους φυσικούς πόρους που αντλούμε. Και τι μπορεί να κάνει η ναυτιλία για να είναι πιο καθαρή, η ασφάλεια στη θάλασσα να βελτιωθεί, όλα αυτά τα λέει θαυμάσια η έκθεση. Ε, μπορούμε να αγωνιστούμε κατά τη πειρατεία και τη ρήπανσης από τα σκάφη. Φυσικά χρειαζόμαστε έρευνα και πόρους από το Connecting Europe Facility. Όλα αυτά τα λέει πάρα πολύ ωραία. Και η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θαλάσσια χωροταξία είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό είναι το κατεξοχήν πραγματικά εργαλείο για να υπάρξει μια βιώσιμη και υφόρος ε, χωροταξία και ένα σχεδιασμό για τη θάλασσα. όχι μόνο στην Ευρώπη, τώρα όλα τα κράτη-μέλη εκπονούν αυτά τα σχέδια, αλλά και διεθνώ, αν καταφέρουμε να το επιβάλλουμε, θα ήταν μία από τι δυνατότητε για να σώσουμε του ωκεανού και να ε, πλαισιώσουμε την αηφόρο ανάπτυξη. Τώρα δεν θέλω να μπω σε όλε τι λεπτομέρειε, είναι πολλά τα καλά και το σημείο 6 για τις λιμενικές εγκαταστάσεις που προλαμβάνουν τη ρήπανση. Ξέρω ότι στη Βαλτική δεν υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις για να αποτρέπουν την ρήπανση όχι μόνο από το διοξίδιο του άνθρακα αλλά και από οξύδια ε, του θείου. Ε, ε, υπάρχει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας που επιβάλλει κάποια μέτρα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και με τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Κύριε Τέιλορ. Yes, thank you, Chair. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, να τη το πείτε παρακαλώ, για αυτό το εξαιρετικό σχέδιο γνωμοδότησης που είναι μέχρι στιγμή ευπρόσδεκτο. Υπάρχουν ωστόσο κάποια θέματα που θα θέλαμε να συμπεριληφθούν στο τελικό, στην τελική γνωμοδότηση και θα υποβάλουμε προτάσεις ή τροπολογίες. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να δούμε τη συμπερίληψη στήριξη για την ΕΜΣΑ και τις αρμοδιότητες της και τα μέτρα για τις ε, εγκαταστάσεις ε, ανοιχτής θάλασσας offshore. Επίσης θα θέλαμε να υπάρξει ισχυρότερη και πιο αποτελεσματική επιβολή της οδηγίας 2005 ε, 35 ε, όσον αφορά την ρήπανση που προέρχεται από τα πλοία. Γιατί ε, δεν επηρεάζονται μόνο οι παράκτητες περιοχές και τα νησιά, οι συνέπειες, από τις συνέπειες μάλλον των κλιματικών αλλαγών, αλλά οι κλιματικές αλλαγές τονίζονται ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τον μαζικό τουρισμό. Θα θέλαμε λοιπόν να τονίσουμε την ιδεολογική συνοχή ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές για την χρηματοδότηση της διακυβέρνησης ε, της θάλασσας και προσβλέπω συνεργασία με τους Κιώδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω ότι ευχαριστώ την εισηγητρία και για την έκθεση και για τη δυνατότητά της να συμπεριλάβει αυτά τα οχτώ στοιχεία με τα πιο σημαντικά θέματα. Να σας πω ότι θα είναι σημαντικό κάποια στιγμή να ταυτοποιήσουμε, να εντοπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν με την υπερβολική ανάπτυξη και αύξηση των ε, εγκαταστάσεων των ε, λιμένων. Δώσαμε προτεραιότητα στους πιο μεγάλους λιμένες και όχι στους πιο αποτελεσματικούς. Αυτό έχει τεράστια αντίκτυπα και στην παράκτια περιοχή και στις λιμανικές, λιμενικές δραστηριότητες, για παράδειγμα τελωνιακές ή υπηρεσίες ασφαλείας. Να επανέλθουμε στις πιο σωστές διαστάσεις, πιο ορθολογικές διαστάσεις των λιμενικών δραστηριοτήτων με καλύτερη και περισσότερη και μεγαλύτερη διανομή, κατανομή μεταξύ των λιμένων. Να μην έχουμε λίγα και τεράστια λιμάνια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια που είναι όλο και μεγαλύτερη, όλο και μεγαλύτερα ενώ ξέρουμε ότι αυτό ε, αποδεικνύεται σήμερα ότι δεν είναι πιο αποτελεσματικό αυτό που είναι απαραίτητο το μεγαλύτερο η αυτοματοποίηση ποιο αντίκτυπο θα έχει στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι κάτι που αξίζει να εξεταστεί. Το αναφέρει η κυρία Μοντέιρο στο σημείο 7. Θα πρέπει όμως να τονιστεί περισσότερο αυτό. Όταν γίνει η πλήρη αυτοματοποίηση των πάντων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα Μπορεί να μην υπάρξουν ανθρώπινα λάθη, γιατί αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε, αλλά μπορεί να υπάρξουν άλλα, άλλου είδους λάθη που θα μας στοιχίσουν πολύ περισσότερο. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να υπάρχει κάποια αναφορά στο Brexit γιατί όλο και περισσότερο μας ανησυχεί αυτό που συμβαίνει με το λιμάνι του Γιβραλτάρ και το στενό του διπυρωτικού διαδρόμου. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρουμε αν θα το πράξει ή όχι, αλλά εν πάση έτσι όπω έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τι συμβαίνει εκεί κάτω, και τι συμβαίνει με αυτό τον διπεριτικό διάδρομο που όλο και εκτείνεται. Και συμφωνώ και υπογραμμίζω την ανάγκη να εξεταστούν και τα θέματα τουρισμού, όχι μόνο στις, τον παράκτιο τουρισμό, αλλά τον τουρισμό κουρασγερόπλιων, ο οποίος είναι όλο και πιο σημαντικός, όλο και μεγαλύτερος, και τα θέματα μόλυσης και ρήπανσης. Ε, ε, για τον ευτροφισμό των θαλασσών μεγαλύτερο αντίκτυπο έχει ο παράκτιος τουρισμός, ο τουρισμός των κουρασγερόπλειων, αλλά και η γεωργική δραστηριότητα. Καλό θα είναι να αναπτυχθεί και το θέμα των εξορρυκτικών δραστηριοτήτων οι οποίες όλο και αναπτύσσονται ε, σε θαλάσσιους πόρους, στη θάλασσα. Και αφού ολοκληρώθηκε αυτή η εξαιρετική μελέτη που ζητήσαμε για το πόσο και κατά πόσο είναι ελκυστικά τα επαγγέλματα των μεταφορών ε, στους νέους και η κυρία Μοντέιρο αναφέρεται αυτό στο σημείο 7. Θα ήθελα να σας ζητήσω, κυρία Πρόεδρε, κάποια στιγμή να γίνει μια σωστή παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή όλων αυτών των θεμάτων. Πράγματι αξίζει η μελέτη αυτή και υπάρχουν ενδιαφέροντα πορίσματα για την ελκυστικότητα των επαγγελμάτων των μεταφορών. Ε, ευχαριστώ, κυρία Γιάλα Σέντερ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Παπακοσταντίνου. Για δύο λεπτά παρακαλώ. <coughs> Ευχαριστώ. Είμαι διευθυντής της Διεθνούς ε, Διακυβέρνησης ε, των Ωκεανών της DG Mare. Ε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Μοντέρο Νταγκηγιάρ και τον κύριο Κάμπο που αρουσίασαν την γνωμοδότηση στα μέλη της Επιτροπής. Είμαι ευτυχής που βλέπω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης καλωσορίζει την ανακοίνωση. Είναι εξαιρετική έκθεση αυτή, πιστεύουμε, και πολύ θερητικό ήταν που ακούσαμε ότι η Κομισιόν ενδιαφέρεται πολύ για όλα αυτά τα ζητήματα, πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά. Είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν και και είπατε εκπρόσωπο εκδίδουν τέτοια είδους δήλωση ε, πολιτικής και αφορά τον ωκεανό, ε, τους ωκεανούς μάλλον. Ε, έχουμε έτσι μια καλή ευκαιρία για να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και να ενισχυθεί η διακυβέρνηση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτό το θέμα, στην διεθνή διαχείριση των ωκεανών, η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος και βασική όθηση για τις κοινέ δράσεις διεθνώς προέρχεται από την Ευρώπη. Ε, αν ε, δούμε λοιπόν ποια είναι η θέση ορισμένων παραδοσιακών μας εταίρων ε, που θέλουν κάπως να μακριθούν, θα δείτε ότι όντως ισχύει αυτό. Ατζέντα 2030 για τους βιώσιμους στόχους, μάλλον στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ε, μπήκε εδώ και επίσης να αναφερθώ στην πρόσφατη διάσκεψη του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για αυτό το θέμα, το που συμμετείχε και η Κομισιόν και το ε, Κοινοβούλιο. Ο σαφής μας στόχος είναι να διατηρήσουμε αυτήν την ε, όθηση και το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή μας στη Μάλτα. 5 και 6 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιλοξενήσει μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς Μεγάλο ορόσημο θα αποτελέσει αυτό, ώστε η πολιτική αυτή να αποσπάσει την προσοχή και του ευρύτερου κοινού. Να τονίσω κάποιες δράσεις που εμπίπτουν σαφώς στην αποκλειστική η κοινή αρμοδιότητα με την Επιτροπή ΕΝΒΙ ή ΤΡΑΝ. Οι εταιρικέ σχέσεις για τους ωκεανούς, ε, βασική δράση της, ε, των ακινοθέντων, όπου προτείνουμε να συναυθούν εταιρικέ σχέσεις με διάφορους χώρε. Στου δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μα. πρέπει να συνεργαστούμε με άλλου μεγάλου φορεί, Αυτό το τονίζει και η κυρία Μοντέρο στη γνωμοδότησή της, στο σχέδιο γνωμοδότησή τη και την ευχαριστώ για αυτό. Επίση, καλωσορίζουμε τη στήριξη τη εισηγήτρια σε σχέση με την προώθηση της θαλάσσια, του θαλάσσιου σχεδιασμού και τη ασφάλεια. Τι εννοούμε, χωροταξία, τη θαλάσσια χωροταξία, το έχουμε κάνει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη και θέλουμε αυτό να γίνει και σε διεθνέ επίπεδο. Η θαλάσσια ασφάλεια επίση αναφέρεται, γιατί κομμάτι τη ατζέντα για τη διακυβέρνηση των ωκεανών έχει το μνηστή και για την παγκόσμια θαλάσσια ασφάλεια, που, ε, την σχετική ατζέντα που υιοθετήθηκε το περασμένο μήνα. Επίση θέλουμε να ανταλλάξουμε διατομεακέ πληροφορίε. Ναι, θα είμαι σύντομο. Ναι, ναι, θα είμαι σύντομο. Τελειώνω. Άκουσα και κάποια σχόλια για το εμπόριο και τον τουρισμό, σημαντικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην ατζέντα για την ε, γαλάζια ανάπτυξη, δημιουργούμε τις προποθέσεις ώστε να παροτρύνουμε την γαλάζια οικονομία. Αυτά λοιπόν περίεκοψα κάπως τις παρατηρήσεις μου, κυρία Πρόεδρε, που μου το ζητήσατε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, με αυτό το ανακοινωθέν έχουμε παρουσιάσει τη φιλοδοξία μας να παίξουμε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των ωκεανών. Έχουμε ήδη στηρίξει και λάβει μάλλον υποστήριξη από το Συμβούλιο που υιοθέτησε τα συμπεράσματά του τον Απρίλιο. Το Συμβούλιο έστειλε πολύ θετικό μήνυμα. Άκουσα απόψε ότι και εσείς στηρίζετε και το Ευρωκοινοβούλιο είναι εταίρος κλειδί για τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας και περνάμε στο επόμενο σημείο. Θυμίζω ότι οι τροπολογίες ε, θα πρέπει να κατατεθούν πριν από τις 14 Ιουλίου στις 10. 14 Ιουλίου στις 10. Θέλετε εκ νέου το λόγο κύριε Πιμβαντερκάμπ. Όχι, απλώ νόμιζα ότι ο εισηγητή ή ο αντικαταστάτη του έχει τον τελευταίο λόγο για να σχολιάσει ε, τις παρατηρήσεις των συναδέλφων πρέπει να πω ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή και με ενδιαφέρον περιμένουμε και τις τροπολογίες. Θα διαβιβάσω τις φιλοφρονήσεις προς την κυρία Μοντέρο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα. Μα εγώ δεν κλείνω, εισηγητής δεν είμαι. Δικαίωμά σα απόλυτο είναι και το διεκδικείτε και το έχετε. Συνεχίζουμε. Προσαρμογή κάποιων άρθρων. Ε, άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρμογή λοιπόν διαφόρων νομικών πράξεων είναι γνωμοδότηση για την Επιτροπή Γιούρη και το λόγο έχει ο κύριος Μάγερ, ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως φαίνεται και από την επικεφαλίδα, είναι ένα θέμα πάρα πολύ νομοτεχνικό αυτό που μας απασχολεί. Και γι' αυτό το λόγο ε, δεν ε, υπάρχει χώρος για πολιτικές, κομματικές ή ιδεολογικές σκοπιμότητες που ορισμένοι επιδιώκουν καμιά φορά. Η Επιτροπή μας νομίζω μπορεί να καλωσορίσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την προσαρμογή ε, στις κατοξιοδότηση και εκτελεστικές ε, εφαρμοστικές πράξεις όπως προβλέπεται και στις συνθήκες της Λισαβόνας. Πολύ σύντομα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της εφαρμοστική Διατάξης μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, δηλαδή να υπάρχουν ενιαίες προδιαγραφές. δεν αλλοιώνουν σε καμία περίπτωση το βασικό κείμενο του δικαίου. Το δεύτερο φορά της κατεξοδότηση πράξης, στο άρθρο 290 ορίζεται αυτό, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, μία κατεξουδότηση πράξη, ούτε αλλάζει, ούτε συμπληρώνει ε, βασικά νομοθετήματα. Άρα η δική μας πρόταση φιλοδοξεί να ρυθμίσει νομικές πράξεις που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο σε 168 περιπτώσεις. Ε, αυτά είναι θέματα της Γιούρη. Για μας 34 ε, έχουν σημασία για την κινητικότητα και την πολιτική των μεταφορών. Περί αυτού πρόκειται συγκεκριμένη νομοδότηση και στις μεταφορές που μπορεί να σας φαίνεται τεχνική απόφαση ε, και όχι πολιτική Ισχύει αυτό. Άρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή να ε, χωρίσει κάποιες αρμοδιότητες, μερικές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι εξασφαλισμένη η νομοθετική διαδικασία. Ουσιαστικά ποια είναι τα τρία πράγματα που μας ενδιαφέρουν και τα θέματα. Πρώτον, η διάρκεια της εκχώρησης αρμοδιοτήτων, μία πενταετία με αυτόματη ανανέωση μετά από έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εννέα μήνες πριν θα πρέπει να καταθέσετε το δεύτερο εξουσιοδότηση για συμπλήρωση της οδηγίας 97 ε, του 70 και του κανονισμού 725 του 2004 και το τρίτο είναι ε, η αλλαγή τεσσάρων οδηγιών. Κάτι άλλο που ήθελα να πω κατόπιν υποδείξεως της Γραμματείας και της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου, έχω συμπεριλάβει στην πρότασή μου τη καλύτερη εναρμόνιση των αιτιολογικών σκέψεων. Θα κάνω άλλες δέκα τροπολογίες λοιπόν για τις αιτιολογικές σκέψεις, έτσι ώστε να ε, το ξέρετε και εσείς σας το λέω από τώρα. Και πιστεύω ότι μπορείτε να εγκρίνετε τις τροπολογίες αυτές και σας παρακαλώ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ποιος έχει τώρα το λόγο. Ο κύριος Κόχ. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής τα είπε πολύ ωραία και τα παρουσίασε. Είναι μάλλον τεχνική έκθεση που αφορά την προσαρμογή στο σύστημα των κατέξουσιοδότης και εφαρμοστικών διατάξεων όπως και άλλες έξι επιτροπές και η Επιτροπή μας γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μάγερ. Ε, είναι πολλά τα καλά σημεία που συμμερίζονται και άλλες επιτροπές και τα στηρίζουν. Ας πούμε, χώριση αρμοδιότητας για ε, της κατεξουσιοδότηση πράξης ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέλει αυτό ε, επαόριστο και το θεωρώ προβληματικό. Γι' αυτό ε, χαίρομαι για την πενταετία που προτείνεται με υποχρέωση έκθεσης για την εκχώρηση αυτή. Επίσης είναι πολύ συνεπής και η συνεργασία και συνεκτική με τις άλλες επιτροπές σε μια τόσο τεχνική έκθεση. Για το λόγο αυτό δεν θα κάνω τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράτος. Eh, Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, το στάκτη γνωμοδότησης καλύτερα, και για τις τροπολογίες τους. Η φιλελεύθερη, θα ακολουθήσει τη γραμμή του Κοινοβουλίου, μια γραμμή που ε, χαράχτηκε το 2013 και απορρέει και από τη Διοργανική Συμφωνία για τη διάρκεια της ισχύω εχώρησης δηλαδή αυτής της δυνατότητας συμφωνούμε για την πενταετία με αυτόματη ανανέωση ε, κατόπιν υποβολής εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και επίσης θέλουμε οι εφαρμοστικές όπως και η κατεξοδότηση πράξης να έχουν την ίδια συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν πρόκειται για διεθνή ε, μέσα και διεθνή συμφωνίες, προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις, αλλά και αυτό με κατεξουσιοδότηση πράξη. Είπε ο εισηγητής ότι οι εξαιρέσεις αυτές έχουν να κάνουν με την ασφάλεια ε, ε της ναυσιπλοείας και όχι μόνο θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο που να το δικαιολογεί. Ας πούμε, ε, η ρήπανση ε, στη θάλασσα ή ε, οι συνθήκες εργασίας των ναυτικών. Πάντως είναι καλή η πρόταση αυτή και ελπίζουμε να συμφωνήσουμε εύκολα και γρήγορα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μαρτίνες κοντά για δύο λεπτά παρακαλώ. Maximum. Το πολύ. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, uh... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του συναδέλφου Αλεχάνδρο Μαρτίνες θα ήθελα να πάρω το λόγο να ευχαριστήσω ε, τον εισηγητή για την παρουσίαση αυτής της γνωμοδότησης. Τα σχόλιά μας θα είναι τεχνικής φύσεως, εξαιρετικά σύντομα, γιατί και η έκθεση αυτή κάθε αυτή είναι τεχνική. Το ακούσαμε αυτό και από τα εξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πήραν το λόγο. Τρία είναι τα στοιχεία που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε. Το πρώτο σχετίζεται με το περιορισμό της δυνατότητας αυτής για μια περίοδο 5 ετών. Και αυτό θα θέλουμε με οριζόντιο τρόπο να ισχύσει για να υπάρχει συνέπεια. Ε, αυτό προτείνεται, αλλά εμείς διαφωνούμε. Γιατί κάθε ανανέωση αυτής της εντολής θα αυξήσει το διοικητικό άχθος και το Κοινοβούλιο έχει πάντοτε το δικαίωμα ανάκλησης και δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε. Με την επαόριστο εντολή. Διατηρείται δηλαδή το δικαίωμα εξέτασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανεξάρτητα από το εάν θα είναι η εντολή επαόριστον. Από τη στιγμή που ανα πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί. Επομένως για μας δεν χρειάζεται η διάρκεια πέντε ετών της εντολής και στη συνέχεια θα ήθελα να σχολιάσω τα, τις τροπολογίες 4, 9, 10 και 37. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι Υπάρχει μια κάποια παρανόηση κατά πάσα πιθανότητα που προκύπτει από, το, από, από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, αυτές οι τροπολογίες αναφέρονται στις διατάξεις που δεν αφορούσαν την ε, κανονιστική διαδικασία με τη διαδικασία εξέτασης. Αυτές οι διατάξεις αφορούν την κανονιστική διαδικασία, άρα δεν έχουν να κάνουν με την άσκηση του κράτους. Δηλαδή, εμείς το θέλουμε αυτό για λόγους διευκρίνησης, για λόγους σαφήνειας και καθαρότητας. Για ορισμένες διατάξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέγραψε το σύνολο του άρθρου στην πρόταση και αυτό το άρθρο περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις που αναφέρονται σε κανονιστικές διαδικασίες με τις οποίες υποτίθεται ότι δεν θα πρέπει να έχει σχέση το εγχείρημα αυτό και η άσκηση αυτή. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω έχει να κάνει με την τροπολογία 3 και την τροπολογία 20. Προτείνεται η αλλαγή της φύσης της νομικής πράξης από, από εκτελεστική να είναι κατεξουσιοδότηση. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμούμε να διατηρηθεί αυτό που προτείνουμε εμείς για την ε, νομοθετική πράξη, γιατί έχουν να κάνουν όλα αυτά με τα ζητήματα εναρμονισμένης ερμηνείας, είναι διαδικαστικά ζητήματα και πιστεύουμε ότι για λόγους κανονιστικούς, διαδικαστικούς, αλλά και για λόγους συνθήκων είναι καλό ε, ο νομικός χαρακτήρας της ε, πράξης να είναι ενιαίος και ομοιόμορφος και εναρμονισμένος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάγερος, εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας. Ε, βέβαια θα κοιτάξουμε αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιμένουμε χαρά τι τροπολογίε σα. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θυμίζω 19 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα και κλεισμένων των θυρών. Με μικρή διακοπή για να σταματήσει η μετάδοση στο διαδίκτυο και να μπορέσει να αποχωρήσει το κοινό και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με την ενημέρωση σχετικά με τους ημερίες διαλόγους και φυσικά όλοι οι βουλευτές μπορούν να παραμείνουν. Allez-y, prenez pas trop votre temps.